Good Χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι, μιλητές, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στην ακρόαση για το μέλλον του Σέγγεν. Το 2016 είχαμε κάνει προηγουμένως αντίστοιχη ακρόαση. Και βλέπετε χρονικά είναι πολύ κοντά τα δύο αυτά. Αυτό τη δείχνει πόσο σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Επίσης αυτό δείχνει πόσο αναπτύχθηκε έκτοτε ε, χώρος Σέγγεν και νομοθετικά και πρακτικά. Όπως γνωρίζετε η διακυβέρνηση του Σέγγεν ε, υφίσταται πιέσεις καθώς έχουμε μεταναστευτική κρίση και ανησυχίες για την ασφάλεια και ορισμένα κράτη-μέλη έχουν διατηρήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για να ανακουφίσουν την κατάσταση πάνω από ένα χρόνο τώρα σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοροφυλακή έχει ενισχύσει την φύλαξη των εξωτερικών μας συνόρων. Έχουν γίνει άλματα στα συστήματα προφόρησης, αλλά απομένουν πολλά ακόμα να γίνουν σε αυτόν τον τομέα με το σύστημα εισόδων-εξόδων, το σύστημα ευρωπαϊκής, ε, το ευρωπαϊκό έγκρισης ε, ταξιδίων και τις αλλαγές στο SIS. Στο μέλλον όλα τα κράτη-μέλη θα ελέγχονται και από ένα νέο μηχανισμό και μια μέθοδο ε, αξιολόγησης ε, κινδύνου και ευάλωτου χαρακτήρα που είναι μια μέτρηση που κάνει η συνοριοφυλακή και η ακτοφυλακή. Η κατάρριξη των ε, συνοριακών ελέγχων είναι από τα πιο απτά και συγκεκριμένα επιτάγματα και κάθε Ευρωπαίο πολίτη μπορεί να το αισθανθεί αυτό και να το εκτιμήσει. Αλλά τώρα έχουμε προβλήματα και προκλήσει εξωτερικά και εσωτερικά, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να είναι ει βάρο αυτού του επιτεύγματο και τη σπουδαία ε, προόδου. Όταν ε, σκεφτόμαστε θέματα ασφαλείας και μετανάστευση. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι στο Συμβούλιο για την πρόοδο σε όλα αυτά τα θέματα. Είναι πιο εύκολο να λέμε ότι, μπορούμε, ότι πρέπει να βρούμε ισορροπημένες λύσεις παρά να το κάνουμε. Αλλά από το 1800 και, το, το, και πιο παλιά κάποιος έλεγε ότι εκείνοι που απεμπολούν την, ασφάλεια, την ελευθερία τους για να έχουν μια στοιχειώδη ασφάλεια δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία ούτε την ασφάλειά τους. Και κινδυνεύουμε να χάσουμε και τα δύο εάν ε, έχουμε ως αντάλλαγμα και τίμημα το ένα στο βωμό του άλλου. Και πιο πρόσφατα το έχουμε δει αυτό στην ιστορία μας. Αυτό ε, που πρέπει να βρούμε είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στην ελεύθερη κυκλοφορία και την ασφάλεια το να ορθώνουμε περισσότερα σύνορα ελέγχους και φραγμούς δεν πρόκειται να βοηθήσει για την ισορροπία. Και πιστεύω ότι η Επιτροπή μας συνέβαλε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για να εξευρεθούν ε, απτές λύσεις, αποτελεσματικές και πρακτικές που να μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη και να βασίζονται και στις αρχές και τις αξίες μας. Ε, ο κούρσα προς τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή όπως είναι ε, ο κανονισμός του Δουβλίνου και τα λοιπά, δεν είναι σωστός τρόπος να εξευρεθεί αυτή η ισορροπία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την προσοχή σας και σε κάποια άλλη εξέλιξη που αφορά το χώρο Σέγγεν. Κυκλοφορούν διάφορες ιδέες να καταργηθούν ε, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έλεγχη στη θάλασσα και στον αέρα και αν κάποια στιγμή αργότερα καταργηθούν, να καταργηθούν ποτέ και στα χερσαία σύνορα. Θέλω να ακούσω την άποψή σας, γιατί αν εγκριθεί αυτή η προσέγγιση θα ήταν μάλλον καινοτομία και μάλλον αφισβητούμενη καινοτομία, έτσι, διότι προς το παρόν είδαμε τι έγινε στη συζήτηση στην Ολομέλεια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο. Πολλοί ομιλητέ στο Κοινοβούλιο έστειλαν ένα χειρό μήνυμα προς το Συμβούλιο κυρίως ότι αυτά που συμβαίνουν είναι αδικία προς τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και παραβίαση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών και των ίδιων τους ε, των υποχρεώσεων. Και είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Η σημερινή ακρόαση λοιπόν έχει ως στόχο να καταγράψει την κατάσταση, να δούμε ποιες είναι οι πρόσφατες εξελίξεις και οι επικείμενες. Και για να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση στο Σέγγεν και πώς αποδίδουν τα μέτρα που ε, ελήφθησαν ή που δεν ελήφθησαν. Και με χαρά επίσης θέλω να πω ότι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας υψηλού επίπεδου ε, εκπρόσωποι από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και το πανεπιστημιακό κόσμο. Θέλουμε να ακούσουμε βεβαίως τα θέματα της απόψης σας και να γίνει και συζήτηση. Δύο λόγια για τη διαδικασία τώρα. Μετά τις δύο πρώτες ενότητες θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Και ε, το τελικό κεφάλαιο, η τελευταία ενότητα, είναι συζήτηση πολιτική υψηλού επίπεδου. Παρακαλώ γνωρίζετε ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο και ε, ε, ηχογραφούνται οι ομιλίες. Αρχίζουμε από το πρώτο πάνελ. Τώρα θέλουμε να δούμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, ιδιαίτερα το σύστημα πληροφόρησης και η εδαφική διάσταση. Έχουμε τον εκτελεστικό διευθυντή της Ιουλίσα, τον διευθύνων Σύμφουλα Κρομ Κάρκοφ, τον δόκτωρα Καρέρα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικών Μελετών και έχουμε και τον Υπουργό, ο οποίος δεν θα μπορέσει να έρθει, ο κύριος Νεγκρέσκου, αλλά ε, ο κύριος Μπογιάντζου τον αντικαθιστά που είναι αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρουμανίας στην μόνιμη ρουμανική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2016 το Τμήμα Πολιτικής για ε, Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές Υποθέσεις ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης ε, για τα ιστορικά σύνορα και τους ελέγχους στο Σέγγεν και ζητήσαμε να μας δώσει μια μελέτη και να μας ενημερώσει ε, το ε, σχετικό τμήμα. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον δόκτωρ Καρέρα. Έχετε 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Ξώτημα μέλη. Είναι πραγματική τιμή για μένα να συμμετέχω εδώ σε αυτή την ακρόαση και να σας παρουσιάσω τα ευρήματα της ε, επικαιροποιημένης ε, μελέτης που έχει κάνει το ΣΕΠΣ για τις τελευταίες ε, εξελίξεις για την κατάσταση στη Σέγγεν. Έχουμε εξετάσει με προσοχή τα τελευταία δύο χρόνια τις εξελίξεις και με τα χαρά να σας δείξω τα ευρήματά μας. Είναι λοιπόν μια μελέτη που έχει ζητήσει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και το Τμήμα Πολιτικής με 19 μέλη, ο Μάρκος Στεφάνσο, επόμενη. Τα ερωτήματα που θέσαμε είναι τρία. Πρώτον, κατά πόσο το σύστημα διακυβέρνηση Έγγεν είναι ανθεκτικό και υπήρξε ανθεκτικό στις κρίσεις. Δεύτερον, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει πέρα ε, της διαμόρφωσης πολιτικής με βάση ε, της ε, κρίσης. Και τρίτον, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά το 2016 έχουμε εντοπίσει και έχουμε εστιάσει την προσοχή μας σε τρεις βασικούς τομείς. Πρώτον, ε, η τρέχουσα κατάσταση ό,τι αφορά την επανεσαγωγή των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων. Δεύτερον, ε, η εσωτερική αστυνομική έλεγχη. Και τρίτον, για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής και μια μικρή επικαιροποίηση σε ό,τι αφορά ε, τα τείχη και τους φράχτες στα σύνορα έχουμε πέντε κράτη-μέλη τα οποία εξακολουθούν να έχουν εσωτερικούς ελέγχους στα σύνορα. Και λέμε ξεκάθαρα στη μελέτη μας ότι έχει τελειώσει ο χρόνος, έχουν παρέλθει οι προθεσμίες με βάση το άρθρο 29 και τώρα τα κράτη-μέλη αυτά θα πρέπει να επανέλθουν στην ε, ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Σέγγεν. Στη μελέτη αναδεικνύουμε ότι πόσο σημαντικό είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει και να ασκήσει πιέσει προ αυτά τα κράτη-μέλη να αιτιολογήσουν κατά πόσο είναι αναλογικά και απαραίτητα τα μέτρα αυτά για του ε, συνοριακού ελέγχου. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ένταση του, αλλά και στον αντίκτυπο που έχουν αυτοί οι έλεγχοι ε, σε όσου του υφίστανται. Μία από τι ε, βασικέ αιτιολογήσει που χρησιμοποιούνται από αυτά τα πέντε κράτη-μέλη είναι ο κίνδυνο δευτερογενών μετακινήσεων. Και εμεί ε, θέτουμε το ερώτημα κατά πόσο αυτό ε, είναι επαρκή αιτιολόγηση για την συνέχιση αυτών των έκτακτων μέτρων. Φαίνεται ότι κάπω είναι θολέ οι διακρίσει και τα η διαφορά μεταξύ των συστήματων ασύλου και εσωτερικής ασφάλειας γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει πραγματικά να δοθεί έμβαση στην ε, μεταγκατάσταση με βάση την μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Είναι λοιπόν ε, σαφές ότι το βασικό ε, θέμα ίσως είναι ότι ακόμα υπάρχει έλλειμμα σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη και τον δίκαιο επιμερισμό των βαρών σε αυτή την περίπτωση επίσης απαιτείται η μεταρρύθμιση του ε, συστήματος ε, ΕΑΣΟ και του ΕΑΣΟ για ε, να έχουμε ένα κατάλληλο σύστημα για όλα τα κρατημέλη, μεταξύ των οποίων και αυτά τα πέντε κρατημέλη που βλέπουν τις δευτερογενείς μετακινήσεις ως πρόβλημα. Η Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό για τροποποίηση του, κώδικα, του συνοριακού κώδικα ΣΕΝΓΕΝ ε, σε ό,τι αφορά την επανεισαγωγή και των εσωτερικών ελέγχων, προτείνεται η χρήση αξιολογήσεων κινδύνου και παρόλα στις ε, σημαντικέ και θετικέ προσπάθειε που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επανέλθουμε στην κανονικότητα, από τη μελέτη μα προκύπτει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα και όχι ε, σε αξιολόγηση κινδύνου. δεν γίνεται να θυσιάσουμε τη Σέγγεν στο βωμό κινδύνων που δεν ξέρουμε κατά πόσο ε, όντως ε, θα λάβουν χώρα. Πρέπει να βασιζόμαστε σε στοιχεία και γεγονότα που ήδη γνωρίζουμε. Γι' αυτό και προτείνουμε να συνδέσουμε αυτή την πρόταση με τον μηχανισμό αξιολόγησης της Σέγγεν που ήδη προβλέπει τη δυνατότητα διαξαγωγή αυτών των αξιολογήσεων στα εσωτερικά σύνορα. Η πρόταση κανονισμού θα μπορούσε πιο επίσημα και τυπικά να διασυνδέσει ε, την ε, να διασυνδεθεί με τον μηχανισμό αξιολόγηση για να δούμε κατά πόσο αυτή η έλεγχη είναι απαραίτητη. Και ε, να υπάρχει και ένα μηχανισμό υποβολή παραπώνων. Αν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που υφίστανται του ελέγχου δουν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Το δεύτερο που εξετάσαμε είναι η εσωτερική αστυνομική έλεγχη. Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση ε, αναλογικών αστυνομικών ελέγχων, σύσταση μάλλον, για, τις, για τους αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους, πιο συγκεκριμένα και για αυτά τα πέντε κρατημέλη. Μία τέτοια σύσταση είναι χρήσιμη, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν μπορούν να ισοδυναμούν με συνοριακούς ελέγχους οι αστυνομικοί έλεγχοι και η σύσταση θα μπορούσε να λάβει υπόψη ε, την τη νομική συγκριτική αξιολόγηση που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην πρόσφατη ε, υπόθεση ΕΣΥ 9 16 για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου και ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για την ε, διενέργεια αυτών των ε, αστυνομικών ελέγχων σε εθνικό επίπεδο για να πληρούνται και οι προδιαγραφές ε, των επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και το ευρύτερο νομικό πλαίσιο. Ένα από τα βασικά στοιχεία εδώ είναι ότι υπάρχει ε, ευελιξία όταν χρησιμοποιούμε αστυνομικούς ελέγχους, αλλά και πάλι δεν είναι ευκρινή τα όρια μεταξύ των ε, δύο. Και όταν έχουμε υπερβολικού αστυνομικού ελέγχου, μπορεί de facto να έχουμε συνοριακού ελέγχου. Από την μελέτη προκύπτει ότι δεν υπάρχει συστηματικός έλεγχος ε, αυτών των ελέγχων και θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα του αριθμού αυτών των ελέγχων και των στατιστικών στοιχείων. Και ποιος ελέγχεται τελικά, ποιος εφίσταται τους ελέγχους και για ποιο λόγο προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα SIS για να παρακολουθούμε την κλίμακα των ε, αστυνομικών ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλής λόγος έχει γίνει για τις βάσεις δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα. Το ερώτημα είναι ποιος έχει πρόσβαση, σε τι και για ποιο λόγο, για ποιο σκοπό. Η αρχή περιορισμού των σκοπών είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν εξετάζουμε και δεν κατονομάζουμε καθώς και ε, ο ιδιωτικό βίος. Και μία από τι βασικέ προκλήσει είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών επιβόλη του νόμου αλλά και μεταξύ των ε, αρχών μετανάστευση και ασύλου που δεν έχουν καμία σχέση με την αστυνομία. Δηλαδή, θα δώσουν πληροφορίε όταν δεν ξέρουν ποιο θα έχει πρόσβαση σε αυτέ. Αυτή η διαλειτουργικότητα λοιπόν τελικά μήπω δημιουργήσει μεγαλύτερη δυσπιστία εντό τη ζώνη Σέγγεν. Αυτό που δεν ε, επιλύεται αυτή τη στιγμή είναι μηχανισμοί ε, υποβολής παραπώνων όταν υπάρχει ε, επαφή με το πρόσωπο αυτό και υπάρχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Αν το πρόσωπο αυτό όμω θεωρήσει ότι δεν είναι με βάση το νομικό πλαίσιο αυτό ο έλεγχο και αν ζητήσει να δει αυτά τα δεδομένα και να δει πού βρίσκονται. Επόμενη διαφάνεια. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή και εμείς την έχουμε εντοπίσει ως μια σημαντική και θετική εξέλιξη υπό το φως ε, της ε, κρίσης αυτής και επισημαίνουμε και τη σημασία της συνοριακής, συνοροφυλακής και ακτοφυλακής για να διατηρήσουμε την επαγγελματική διάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τους ε, συνοριακούς ελέγχους και την διαχείριση των συνόρων. Είδαμε πως η παρουσία της Frontex διασφαλίζει ότι την αξιολόγηση ομοτήμων με τους εθνικούς ε, αξιωματούχους που είναι βασικό στοιχείο για την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων. Ε, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις ε, που αφορούν την εξάρτηση του οργανισμού από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ακόμα μεγάλος βαθμός εξάρτησης της νοριαφιλικής και ακτοφυλακής από τα κράτη-μέλη. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και κατακαιρματισμένο πλαίσιο παραγόντων σε εσωτερικό επίπεδο. Οπότε πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ ό,τι αφορά το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη νέα Frontex. Μία σειρά ζητημάτων θα μπορούσε επίση να αναλάβει που αφορούν τον μηχανισμό υποβολή παραπώνων τη Frontex, που ακόμα δεν είναι ανεξάρτητο. Ίσως θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερε προσπάθειε για να διασφαλίσουμε ότι, τα, ότι η αρχή θεμελιωδών δικαιωμάτων θα έχει περισσότερη ανεξαρτησία και δυνατότητες να ελέγχει ε, τις ε, επιχειρήσεις της Frontex και κατά πόσο πληρούν και συμμορφούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το τελευταίο που κοιτάσαμε είναι τα ε, σύνορα, τα τείχη και φράχτες στα σύνορα. Και είδαμε ένα ντόμινο ουσιαστικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτή την άποψη. αυτό γύρει ζητήματα συμβατότητας ε, αυτών των τυχών και φραχτών και με τις ευρωπαϊκές αξίες που ανέφερε πολύ σωστά ο Πρόεδρος, αλλά ε, και με τον SIS, τον κώδικα SIS και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γιατί βλέπουμε ότι έτσι επιτρέπονται παράνομες ε, πρακτικές σε ορισμένες χώρες, και εμείς συζητούμε να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτό το θέμα, γιατί ενδεχομένω να υπονομεύσει την νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε αυτό το τομέα. Κλείνοντα. συστήνουμε η λήψη αποφάσεων με βάση της κρίσης ως επιχείρημα να μην χρησιμοποιείται πια ιδίως από Υπουργεία Εσωτερικών, για να ε, αναστείλουν ε, την, ε, τον εξευρωπαϊσμό ή την λισαβονοποίηση της Σέγγεν. Και εδώ είναι σημαντική και η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Όμως δεν μπορούμε στο όνομα των κρίσεων να θυσιάσουμε αυτά που έχουμε ήδη ως πρότυπα που είναι μοναδικά. Εμείς συμπεραίνουμε ότι η Σέγγεν όντως είναι εύρωστη και έχει ανθεκτικότητα στις κρίσεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η Σέγγεν, είναι το κεκτημένο ε, ως προς το άσυλο. Πρέπει να απομακρυνθούμε λοιπόν από τον υφιστάμενο ε, κανονισμό του Δουβλίνου που ακόμα βασίζεται σε άδικο επιμέμου ευθυνών και υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να επιλύσουν τις δευτερογενείς ε, μετακινήσεις, ε, καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου. Θα μπορούσε να συνδράμει κράτη-μέλη όπως η Αυστρία, που από ό,τι φαίνεται ε, έχει προβλήματα με τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καρέρα, που τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Μποϊαντζού, που είναι αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος για τη Ρουμανία, για να μας μιλήσει για την εδαφική εμβέλεια ε, του χώρου Σέγγεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Ε, με μεγάλη χαρά και τιμή ήρθα εδώ για να σας μιλήσω σήμερα εκ μέρους του αναπληρωτή Υπουργού του κύριου Νεμπρέσκου για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ήθελε πάρα πολύ να έρθει εδώ σήμερα, αλλά τελικά ε, παρότι, δεν, δεν, ήθελε δεν μπορούσε και έπρεπε να παραμείνει στη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ για αυτή την ακρόαση και σας ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα για τη χώρα μου. Ο χώρος Σέγγεν είναι βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η Ρουμανία ε, έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει και να ενισχύσει το χώρο αυτό. Μιλάμε πολύ αυτές τις μέρες για το μέλλον της Ευρώπης και αυτό συνδέεται με τις προοπτικές ε, μιας ε, ε, λειτουργούσας και αποτελεσματικής περιοχής Σέγγεν. Είναι ένα από τα project το Σέγγεν που δείχνει την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη διατηρήσουμε, κρατώντας την ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη κυκλοφορία και την ασφάλεια. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο όταν συντονίζουμε το πλαίσιο Σέγγεν που θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η χώρα μου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 είναι ένας εταίρος αξιόπιστος ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για το κεκτημένο Σέγγεν και για την εφαρμογή του και υιοθετεί μέτρα για να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα υψηλότερα πρότυπα. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σας μιλήσω για τα βασικά μέτρα και της Πρωτοβουλία της Ρουμανίας με άμεση επίπτωση στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στη μετανάστευση και τη συνεισφορά μας στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση του Σέγγεν και την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία μαζί με τα άλλα κράτη-μέλη ε, εμπλέκεται στις συζητήσεις ενεργά για τη βελτίωση της διακυβέρνησης του χώρου Σέγγεν. Ο τελικός στόχος είναι να ξαναρχίσουμε, ε, να επιτρέψουμε στο Σέγγεν να λειτουργεί πλήρως ε, προς όφελο όλων των πολιτών και της ασφάλειας συμμετέχει η Ρουμανία με εμπειρογνώμονε ε, σε επιτόπιε επισκέψει αξιολόγηση, σε άλλα κράτη-μέλη, σε όλου του τομεί αξιολόγηση του χώρου Σέγγεν. Ε, σε ό,τι αφορά την συνεισφορά σε εμπειρογνώμονε, μαζί με την Πορτογαλία το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν από τα καλύτερα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά αυτέ τι επιδόσει. Άλλε, επίση, ε, υιοθετήσαμε τον κανονισμό 454 για, το, για την εμβέλεια της, ε, του Σέγγεν. Ε, θέλουμε συστηματικούς ελέγχους, χωρίς εξαιρέσει. Ε, είναι απαραίτητο μέτρο για να υπάρχει ε, αυστηρότατος έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα. Είμαστε από τα πρώτα κρατημέλη που ε, εφαρμόσαμε επιτυχά το σύστημα Eurosource. συμμετέχουμε με πληροφορίες στις επιχειρησιακές δραστηριότητε, για την λαθρομετανάστευση ε, περιστατικά σε διαλέψεις στα σύνορα. Σε ό,τι αφορά το μελλοντικό πλαίσιο ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε υπέρ τη υιοθέτηση και εφαρμογή ε, του πακέτου για τα έξυπνα σύνορα, το σύστημα εσόδου-εξόδου, το σύστημα ε, αξιολόγηση ε, για του ταξιδιώτε κτλ. Το, και, καθώς και το EU LISA. Ε, παράλληλα, ω τμήμα των προσπαθειών τη, η Ρουμάνια ήταν ε, το δεύτερο κρατό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γαλλία που έχει δημιουργήσει ένα εθνικό PNR. Έχουμε δηλαδή μία μονάδα που ασχολείται με τι πληροφορίε για του ε, επιβάτε και του ταξιδιώτε. Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε και να προσαρμόσουμε το νομικό πλαίσιο με βάση τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ούτως ώστε να μην υπάρχουν κενά στην αρχιτεκτονική δομή της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στις κοινέ προσπάθειές μας, τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης είναι πιο ισχυρά και πιο ασφαλή σήμερα. Είναι προφανές ότι με συνεργασία μπορούμε να έχουμε και ασφάλεια και ελευθερία κυκλοφορία στα πλαίσια της κρίσης μετανάστευσης, η Ρουμανία έδειξε την διάθεσή της να επιμεριστεί τις ε, ευθύνες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν το 2015, η Ρουμανία έχει μια δέσμευση να λάβει 4.180 ε, ανθρώπους, να υποδεχθεί δηλαδή και να να μεταφέρει ε, με το πρόγραμμα νόμιμης ε, ε, κατάστασης 995 Σύριους από την Ιταλία και Ιταλία. Μέχρι στιγμής έχουμε δεχτεί 728 από την Ιταλία και Ελλάδα ε, με βάση την ποσόστοση 2.182. Ε, είμαστε από τα πιο δεσμευμένα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την ε, κατάσταση, έχουμε δεχθεί το 1743 από την Τουρκία. Το 2017 και 2018 θα συμμετέχουμε στις προσπάθειες κατάσταση. Τώρα, επίσης απέναντι ε, στου οργανισμού, έχουμε δείξει πολύ θετική στάση. Το 2016 και το 2017 η Ρουμανία ε, είχαμε, είχε πολύ σημαντικέ συνεισφορέ στι αποστολέ Frontex ε, με αμπειρογνώμονε και εξοπλισμό που διαθέσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το 2018 ε, θα συνεχίσουμε την, να συνεισφέρουμε συμμετέχοντα με προσωπικό και εξοπλισμό στι ε, στις στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με σεβασμό των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει προ αυτήν την κατεύθυνση με συνεπή τρόπο για να υποστήριζουμε τις δράσεις της, ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου ε, Υποστήριξη ε, για το Άσυλο. Έχουμε συνεισφέρει στην εργασία της ΕΑΣΟ, συμμετέχοντας με πυρογνώμονε στην ΕΑΣΟ, στις αποστολές ε, στην Ελλάδα, Ιταλία και Βουλγαρία ανάμεσα στο 2014 και το 2017, σε αυτά τα έτη δηλαδή. Φέτος η Ρουμανία είναι διεθυμένη να συμμετέχει ε, στις επιχειρήσεις του ε, ΕΑΣΟ στην Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία. για τα θέματα ε, των ευάλωτων ανθρώπων, ε, πληροφορίες για την ε, επανεγκατάσταση και, για, και βοήθεια για την εξέταση των αιτήσεων για αυτό που, ζητούν διεθνή προστασία. Τώρα, για να αντιμετωπίσουμε τις τρομοκρατικές απειλές, εμείς έχουμε υποστήξει όλα τα μέτρα που έχουν σαν σκοπό να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία για την άμυνα των, και προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και να συνεργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, καθώς και με τρίτες χώρες. Ε, αυτό το έχουν αγνωρίσει όλοι οι εταίροι μας και έχουν τονίσει τη θαυμάσια συνεργασία με τι Ρουμανικέ Αρχές για να καταπολεμήσουμε ε, το πρόβλημα των ε, ξένων μαχητών. Πού βρισκόμαστε σήμερα η συμμετοχή της ε, Ρουμανίας σε όλα τα θέματα που αφορούν την ε, ασφάλεια δείχνει την προσθέμενη αξία για την ε, ενδυνάμωση του χώρου Σέγγεν και της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανία είναι ένας εταίρος που βοηθάει και στηρίζει την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν πάντα δήλωνε ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία πληρούν όλα τα κριτήρια για να προσχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις υποστηρίζει. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω ότι το αναγνωρίζει αυτό ε, το Κοινοβούλιο ότι είμαστε έτοιμοι δηλαδή και εμείς και η Βουλγαρία και ελπίζω να μας υποστηρίξετε και περαιτέρω σε αυτό το διάλογο με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ε, η Κομισιόν τόνισε την ανάγκη να εντάξουμε πλήρως την Βουλγαρία και την Ρουμανία στο Σέγγεν γιατί μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να έχουμε μια ισχυρότερη περιοχή Σέγγεν. Όμως δεν υπάρχει ομοφωνία ακόμα στο Συμβούλιο για την ε, προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας παρά το γεγονός ότι πληρούμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ε, σε διαδοχικέ αξιολογίες που έχουν γίνει. Θα, αν προσχωρήσουμε πλήρω, ε, θα συνεισφέρουμε στο χώρο Σέγγεν. Έτσι πρέπει να, να θεωρηθεί αυτή η συμμετοχή μα, σε μια εποχή που αμφισβητείται το Σέγγεν όλο και περισσότερο. Και θα είναι και πολιτικό ε, μήνυμα για την βιωσιμότητα του project που λέγεται Σέγγεν. Η Ρουμανία παραμένει σήμερα ένας αξιόπιστος εταίρος ε, για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος. Οποιοδήποτε άλλο σενάριο είναι αντίθετο στις φιλοδοξίες, ε, τις αξίες και τις πεπιθήσεις μας, ε, πεπιθήσεις που πάντα και αξίες που πάντα προωθεί η χώρα μας. Εμείς στα πλαίσια της αλληλεγγύης και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε να δρούμε έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα, καμία ρογμή στην ασφάλεια και είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν την διεύρυνση του Σέγγεν. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο με όλα τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να έχουμε μια θετική απόφαση για το θέμα αυτό και είμαστε προσιλωμένοι στις ε, ευρωπαϊκές αξίες και ε, βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου ε, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε που Μας παρουσιάσετε τα, τις πρόσφατες εξέλιξεις στο θέμα αυτό. Τώρα για τα συστήματα ενημέρωσης και πληροφοριών θα, το SIS θα δώσω το λόγο στον κύριο ε, Γκάρκοφ από την Λίσσα. Ε, ευχαριστώ αξιότιμοι κύριε και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς ε, θα ήθελα να παραθέσω κάτι που είπε ο πριν από 20 χρόνια και πλέον. Ότι είναι μόνο μία Ευρώπη και την είδα εγώ από το παράθυρο του αεροπλάνου. Τι σημαίνει αυτό για το Σέγγεν. Αυτό αφορά ε, ε, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει μεγαλύτερο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ενότητας από το Σέγγενα. Δεν είναι μόνο θεμελιώδης πυλώνας, είναι και ένα σύστημα φιλόδοξο, σύστημα συνεργασίας και αλληλεγγύης ε, μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και την ενιαία αγορά. Οι κανονικοί πολίτες, οι συνήθεις πολίτες έχουν καταλάβει ε, τι ακριβώς είναι το Σέγγεν. Είναι περίπλοκο ε, νομοθετικά και διοικητικά και τεχνολογικά, αλλά ε, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία ενό χώρου χωρίς σύνορα. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι σημαντική ως επιτεύγμα της ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με τις πρόσφατες στατιστικές, έχει τετραπλασιαστεί η κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εξωτερική μετανάστευση. Θα πρέπει να ασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό της Ευρώπης. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ε, πλεονέκτημα και σε ε, εποχές ε, οικονομικής δυσκολίας ε, είναι πολύ σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε όλο το εργατικό δυναμικό όλες οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σύνορα να είναι ανοιχτά, να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά ταυτόχρονα και ασφαλή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Σέγγεν έχει γνωρίσει μια μεταμόρφωση ριζική. Πρώτον, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ε, σύγκληση μεταξύ της διαχείρισης της μετανάστευσης των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας. Δεν υπάρχουν ακόμα πλέον ε, διαχωριστικές γραμμές. Ταυτόχρονα, η κανονική λειτουργία του Σέγγεν σήμερα εξαρτάται απολύτω από την πληροφορία και την ανταλλαγή των πληροφοριών. Άρα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να λειτουργήσει σωστά σήμερα ο χώρος Σέγγεν και στο μέλλον είναι ε, τα μεγάλα συστήματα ε, υπολογιστών και πληροφορικής που υπάρχουν πάντα στην Ευρώπη. Το SIS, σύστημα πληροφόρηση Schengen, ήταν το πρώτο αντισταθμιστικό ε, μέτρο για την άρση των εσωτερικών συνόρων. Και σήμερα παραμένει αυτό. Σήμερα το SIS είναι το πιο ισχυρό σύστημα πληροφορικής στην Ευρώπη που χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την επιβολή του νόμου και του συνοριακούς ελέγχους. Τα στοιχεία προσωρινά για το 2017 δείχνουν ότι το SIS 2 έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 5 δισεκατομμύρια φορές από όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή ε, μία, ένα δισεκατομμύριο περισσότερες φορές από ότι ε, το 2016. Αυτή η αύξηση λοιπόν της ε, χρήσης δείχνει ε, και τις επισκέψεις το 2017, πάλι ε, στοιχεία προσωρινά δείχνουν ότι τα hits αυξήθηκαν κατά 20% και σε αριθμούς απόλυτους αυτό σημαίνει πάνω από 240.000 ε, hits για πρόσωπα. Με τις νέες δυνατότητες θα έχουμε και προστιθέμενη αξία για την εσωτερική διαχείριση των συνόρων. με πλήρη βιομετρικά στοιχεία και ελέγχους για τις εισόδους βάσει ε, των θεωρήσεων Σέγγεν. Πάνω από 52 εκατομμύρια αιτήσει έχουμε και 44 εκατομμύρια ε, δακτυλικά αποτυπώματα. Στη Eurodac είναι 6,5 εκατομμύρια ε, τα αποτυπώματα που είναι αποκοινωμένα. Τι δείχνει το σύστημα σήμερα, ότι θα πρέπει να εξελιχθεί για να ανταποκρίνεται στο μέλλον ε, και στους στόχους της ε, σχετικής πολιτικής. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη πρόοδος ακόμα προς την ολοκλήρωση των προτάσεων αναδιατύπωσης του SIS2 και του Eurodac και στα κράτη-μέλη και στο Σέγγεν. Αυτό θα βοηθήσει ως ανταλλαγή ε, πληροφοριών σε ένα σύστημα για μετανάστευση και επιβολή του νόμου. Και αντίστοιχα για τις θεωρήσεις Σέγγεν αργότερα του έτους. Έχουμε επίσης ε, και τον έλεγχο εισόδων και εξόδων. Αυτά τα δύο συστήματα θα συνεισφέρουν ε, άμεσα και σε ένα έλεγχο για προέγκριση θεώρησης ε, διαβατηρίου για πολίτες τρίτων χωρών θα βοηθήσει την ασφάλεια ε, στο χώρο Σέγγεν και είναι θετική η απόκριση που έχει δοθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν και να έχουν πρόσβαση στο Σέγγεν με στοιχεία και δεδομένα υψηλή ποιότητα. Επίση, για να υπάρχει καλή λειτουργία και με διαφάνεια του Σέγγεν στο μέλλον, θα πρέπει να σπάσουν τα, ε, οι φραγμοί που υπάρχουν ακόμα. Ε, ε, έγινε μια πρόσφατη ε, πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων προφορική. Είναι σημαντικό αυτό. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να επιτελέσει σημαντική και ταχεία πρόοδο για να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη από το υπάρχον και νέα συστήματα, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, βέβαια σεβόμενη πάντα τον περιορισμό των στόχων η διαλειτουργικότητα δεν έχει στόχο να ε, έχουμε διπλά συστήματα ε, ενημέρωσης, αλλά ε, πιο καλή διαχείριση. Θέλουμε έξυπνα συστήματα, διαλειτουργικά για το μέλλον και αυτό θα είναι ο ακρογωνιαίος λήθος για το Σέγγεν τον επόμενο αιώνα. Κυρίες και κύριοι, η αποστολή της ε, Γιουλίζα είναι να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη ε, στην προσπάθειά τους να κάνουν την Ευρώπη πιο ασφαλή. Από την ίδρυσή μας, ο οργανισμός μας είναι σημαντικό θεμέλιο του Σέγγεν και καθαρό συνεισφορέα στην καλή λειτουργία του. Τα επόμενα έτη η Γιουλίζα θα εξακολουθήσει να ε, επιτελεί το έργο της, την αποστολή της και το ρόλο της. Ταυτόχρονα και με τις δράσεις αυτές θα συμμορφωθούμε πλήρως με τις αρχές προστασίας προσωπικής ιδιωτικής σφαίρας, δεδομένων και ε, πληροφοριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάρκοφ. Αρχίζει τώρα η συζήτηση ε, για τους βουλευτές που ζητούν το λόγο. Η κυρία Γκραπίνη πρώτη. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για την διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, στα τέλη της περασμένης χρονιάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε ψήφισμα με το οποίο ε, ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξει την πρόσβαση της Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν και της Βουλγαρίας. Όχι επειδή είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία, αλλά επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης και ένταξης. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καρέρα για την πολύ καλή παρουσίαση και να τον ρωτήσω το εξής. Είπατε, κύριε Καρέρα, ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε γεγονότα και στοιχεία και όχι στον κίνδυνο. Εγώ προέρχομαι από το επιχειρηματικό περιβάλλον και αν προσπαθούσα να πάρω μία ε, απόφαση βάσει του ρίσκου, βάσει του κινδύνου, ίσως να μην ήμουν σε θέση να φτιάξω μια επιχείρηση. Πράγματι δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τους κινδύνους, όμως μπορώ να σας πω ότι στη Ρουμανία ο κίνδυνος ε, μιας ε, τρομοκρατικής επίθεσης και άλλων ε, αρνητικών φαινομένων που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μικρός. Πολύ μικρότερος λοιπόν στη Ρουμανία σε σχέση με άλλες χώρες που αντιτίθενται στην ένταξη της Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν. Εδώ και δέκα χρόνια λοιπόν είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ ψηλό ποσοστό στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρουμανία, το οποίο τώρα έχει αρχίσει να μειώνεται. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ε, μια ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί έχουν, έχει αυξηθεί, έχει αναπτυχθεί ο ευρωσκεπτικισμός, δείτε τι συνέβη με τον Brexit. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς επιθυμούμε και επιδιώκουμε να πετύχουμε με τις πολιτικές μας. Πολλοί με ρωτούν γιατί δεν έχουμε ακόμα ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν, κάτι το οποίο επηρεάζει τόσους πολλούς πολίτες. Τόσους πολλούς πολίτες. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είμαστε ακόμα μέλος. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι συνομοθέτε θα πρέπει να λάβουν από κοινού μια απόφαση. Και νομίζω ότι η δημοκρατία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή, καθώ ε, και η αρχή τη πλειοψηφία. Δυστυχώ δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Καλό είναι λοιπόν να μείνετε στο ένα λεπτό. Ο κύριος Κοέλιο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, Δ. Καρέρα. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Αυτή είναι και η εκτίμηση του Κοινοβουλίου, ότι η Σέγγεν ε, θα είναι μέλος της, μέρος της λύσης, δεν είναι μέρος του προβλήματος. Και επισημάνατε πολύ σωστά και ε, τη σημασία του κανονισμού του Δουβλίνου και τις ευθύνες που διερρύπτονται. Όμως έχω ακόμα δύο ερωτήματα. Μιλήσατε για την διασύνδεση μεταξύ του μηχανισμού αξιολόγησης Σέγγεν και ε, τους ελέγχους και των ελέγχων των συνεργειακών. Ε, πώς ακριβώς βλέπετε αυτή τη ε, διασύνδεση. Και δεύτερον, μιλήσατε για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διακυβέρνηση σε επίπεδο Σέγγεν. Ποια είναι η πρόταση διεύρυνση και να επιτρέψουμε την ε, συνέχιση αυτών των συνεργειακών ελέγχων ή νομίζετε ότι κάτι θετικό μπορεί να προκύψει. Για τη Ρουμανία να πω ότι συμφωνώ σας ασκήσαμε πιέσεις, κάνατε αυτό που έπρεπε να κάνετε, Ρουμανία και Βουλγαρία, και οι ε, εμπειρογνώμονες επιβεβαιώνουν ότι είχατε δίκιο, δεν σας έχει προδώσει το Κοινοβούλιο, αλλά όπως είπατε το πρόβλημα είναι η ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή την Προεδρία έχει η Βουλγαρία στο Συμβούλιο και το ζητούμε από την Βουλγαρία να ε, προχωρήσει σε ορισμένους φακέλους ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του SIS. Υπάρχουν ε, θετικά σημάδια ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος και να προσχωρήσουν όντω αυτές οι δύο χώρες ε, στον, στο χώρο Σέγγεν μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Χαλάο. Ευχαριστώ πολύ. μία ερώτηση και ένα σχόλιο προς τον κύριο Καρέρα. Είπατε ότι πρέπει να έχουμε ένα σωστό κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρώπη και ένας αυτόματος μηχανισμός μετακατάστασης θα ε, μπορούσε να άρει αυτό το φαινόμενο των δευτερογενών μετακινήσεων. Όμως αυτό είναι ρεαλιστικό γιατί έχουμε δευτερογενείς μετακινήσεις, γιατί κάποια κράτη-μέλη είναι πιο ελκυστικά από ό,τι άλλα από την πλευρά του ε, του άσυλο. Ακόμα και αν υπάρχει λοιπόν αυτόματη μετακατάσταση ενός προσώπου σε ένα κράτος μέλος που δεν θέλει να πάει, θα φύγουν από εκεί και θα πάνε ε, εκεί που θέλουν, εκμεταλλευόμενοι και ε, τα ανοιχτά σύνορα. Ενδεχομένως λοιπόν να έχουμε πολύ λίγες εναλλακτικές λύσεις ε, αντί των ε, εσωτερικών μητρικών ελέγχων αν θέλουμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο δευτερογενών μετακινήσεων. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και φαντάζομαι εννοείται ότι θα πρέπει να θέσουν τέλο στου εσωτερικού ελέγχου στα σύνορα το στομότερο δυνατόν. Συμφωνείτε όμως ότι η επανεισαγωγή των ε, συνοριακών ελέγχων ήρθε ως απάντηση σε απρόβλεπτες και έκτακτες καταστάσεις. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο αυτά τα πέντε κρατημέλη κάνουν ε, για πλάκα. Το κάνουν επειδή πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικά και υπαρκτά προβλήματα. Ευχαριστώ. Κύριος Ράντεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η διεύρυνση του χώρου Σέγγεν για να συμπεριλάβει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ήταν αντικείμενο πολλών συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ' επανάληψη είπε ότι οι χώρες ε, εκπληρώνουν όλα τα τεχνικά κριτήρια που είναι τα μόνα νομικά κριτήρια και η μόνη προϋπόθεση για την προσχώρησή τους. Η συμμορφούνται με την νομοθεσία Schengen, χρησιμοποιούμε το SIS, το SIS δηλαδή, και το Συμβούλιο στην αρχή της χρονιάς υιοθέτησε μία απόφαση να επιτρέψει πρόσβαση 100% εμείς αναγνωρίζουμε την, ε, τις θεωρήσεις Schengen, ε, χρησιμοποιούμε το ETIAS. Επομένως, η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι de facto μέλη του χώρου Schengen. Αλλά εξαιτία κάποιων κρατών μελών και των αντιρρήσεων που φέρουν, δεν είμαστε και τυπικά μέλη. Είναι θλιβερό που επιτρέπουμε στις πολιτικές και μικροπολιτικές να παρεμποδίσουν ε, και να εμποδίσουν να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μία αποστολή στη Βουλγαρία και οι ευρωβουλευτές μπόρεσαν να δουν δύο ισόμασοι πώς ε, τα βουλγαρικά ε, σύνορα προστατεύονται με ελέγχους και πώς η Βουλγαρία ε, προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα. Φέτος θα έπρεπε κανονικά να είμαστε ικανοποιημένοι και να, και να επωφεληθούμε από την διεύρυνση του Σέγγεν ε, και την ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ευχαριστώ κύριε Βίξτρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε σε αυτή την ακρόαση. Είναι η χρυσή ευκαιρία για μας ε, για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Είμαι εισηγητής για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Καρέρα ότι ως αποτέλεσμα του αποτυχημένου συστήματος κοινού ασύλου ε, ζούμε σήμερα την κατάσταση που ζούμε εδώ και καιρό. Σήμερα το απόγευμα Διάβαζα την αξιολόγηση της ε, Σουηδίας ε, και εμείς βλέπουμε πώς τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν την ευκαιρία για να προκαλέσουν σύγχυση ανάμεσα στο άσυλο και την ασφάλεια. Με συνοριακούς ελέγχους καταρχήν, κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης, μετά ε, άρχισαν να μιλάνε για ασφάλεια. Τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε όλα αυτά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα νέο σύστημα Δουβλίνου που θα βασίζεται σε μόνιμες κατανομές. Δεν μιλάμε για ε, μετεγκατάσταση, αλλά για εγκατάσταση, όπου όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και αναλαμβάνουν το βάρος που τους αναλογεί. Ε, την ε, έννοια πέντε ε, μεγάλες ομάδες, το 75% των ε, μελών εδώ του, του οίκου μας, ε, συμφωνούν. Εγώ ήμουν ε, σε 23 συνεδριάσεις ε, σκιωδών εισηγητών. Άρα το Συμβούλιο είναι εξαφανισμένο. Δεν υπάρχει δηλαδή διαπραγματευτής, δεν υπάρχει κάποιος απέναντί μας για να συζητήσουμε. Καλό τους υπουργούς εσωτερικών να μην ασκούν πολιτική με βάση την κρίση πια. Εδώ εμεί στο Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, αλλά δεν έχουμε συνομιλητή. Μπορείτε να μα δώσετε λίγα περισσότερα επιχειρήματα για τι επερχόμενε μάχε με το Συμβούλιο. Σα παρακαλώ, κύριε Καρέρα. Ο κύριο Δία Ντεμέρα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του τρει ε, εισηγητέ και για τα σχόλιά τους. Το μέλλον θα πρέπει να μας βρει δυνατούς η ελεύθερη διέλευση θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η έλεγχη θα πρέπει να είναι προσωρινή. Πολύ με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία να είναι μέλη 100%. Γιατί νομίζω ότι πληρούν όλα τα κριτήρια που έχουμε βάλει. Τρίτο σχόλιο για τον Ιουλίσσα. Το ΒΙΣ, το SIS και το Eurodac, ε, το σύστημα εισόδου-εξόδου και το ETIAS. Όμως μας λείπει το ΕΚΡΙΣ και το PNR. Το EU, η e Μετά τις νομοθετικές προτάσεις για τη λειτουργικότητα που μας ανή, ε, ο Επίτροπος King, ε, πλέον θα υπάρχει πληρότητα, ε, θα έχουμε όλα τα στοιχεία για την ασφάλεια. Ευχαριστώ, κύριο Βαλέρο. Η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά, αφού μπορώ. Στη Σουηδία, ε, μέχρι το 1994 από τη δεκαετία του 1980 μέχρι το 1994 ε, υπάρχει μια ένωση σε όλη τη Σκανδιναβία. Δεν χρειάζεται κανείς ε, για διαβατήριο για να ταξιδέψει από μια σκανδιναβική χώρα σε μια άλλη. Εμείς από το 1974 ε, ταξιδεύουμε ελεύθερα χωρίς διαβατήρια. δεν υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι. Και αυτό ίσχυε μέχρι πρότινος. Τώρα όμως άλλαξε η κατάσταση κλείσαμε τα σύνορα ε, για ένα χρονικό διάστημα όταν ερχόταν κανείς από την ε, Κοπεχάγη στο Μάλμε ε, μια, ένα δρόμο ας πούμε, που παίρνω πολύ συχνά βλέπω ότι υπάρχουν συχνά έλεγχοι. Αρχικά ελέγχαν τα διαβατήρια. Έπρεπε μάλιστα να κατέβουμε και από τα τρένα, ας πούμε, στην Σουηδική πλευρά. Είχαν, είχαμε και αστυνομικού ελέγχους. Τώρα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Πάντα πρέπει να δείχνει το διαβατήριό σου στους αστυνομικούς όταν φτάνει στη Σουηδία. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία. Υπάρχουν και άλλοι ε, έλεγχοι. Όταν ε, ταξιδεύω στη Στοκχόλμη και κατεβαίνω εκεί στο τρένο, εγώ δεν θυμάμαι επί χρόνια να δείχνω ποτέ το διαβατήριό μου. Και τώρα ξαφνικά πάμε στο Στρασβούργο, α πούμε, ε, στη Γαλλία ε, πάμε μία φορά το μήνα και όταν κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο θα πρέπει να περνάμε από τον έλεγχο των διαβατηρίων. Όμως όταν φτάσω από τη Φραγκφούρτη με αυτοκίνητο και πολλοί ε, ευρωβουλευτές πάνε από τη Φραγκφούρτη στο Στρασβούργο δεν υπάρχει έλεγχος, κανένας έλεγχος εκεί. Τι κάνουμε λοιπόν με του συνοριακού ελέγχου. Υπάρχουν δηλαδή ε, συνοριακοί έλεγχοι, αλλά μόνο σε συγκεκριμένε περιοχέ. Δεν είναι λίγο περίεργο, δεν είναι λίγο αστείο. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, είπα διάφορα, ξεχάστηκα λιγάκι, αλλά πραγματικά διρωτώ με τι συμβαίνει. Υπάρχουν τώρα νέες απειλές. Τότε πρέπει να δούμε και τις συνέπειες. Κύριος Ευχαριστώ πολύ. Είμαι μηχανικός και πρακτικός άνθρωπος και μου αρέσουν τα στοιχεία και ευχαριστώ τον κύριο Καρέρα που μας είπε αριθμητικά στοιχεία και ε, συζητούμε για την ένταξη Ρουμανίας και Βουλγαρίας στο Σέγγεν. Κάποια άλλα στοιχεία τα είπαν και οι συνάδελφοι, θα ήθελα όμως να επιμείνω. Είπατε ότι πέντε κράτη-μέλη συν η Γαλλία πρέπει να διατηρήσουν τους συνοριακούς ελέγχους, να καταργήσουν μάλλον. Ε, το συζητούμε και στην Επιτροπή για την Τρομοκρατία, την ειδική που έχουμε συστήσει. Και φυσικά θα πρέπει να τερματιστούν τώρα αυτοί οι έλεγχοι και να επανέλθει η ενότητα στο χώρο Σέγγεν. Αφήστε δε που η Ρουμανία και η Βουλγαρία πληρούν όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν πολιτική απόφαση και η Βουλγαρική ε, Προεδρία, η Αυστριακή, το αργότερο η Ρουμανική Προεδρία θα πρέπει να κάνουν την πρόταση για την ένταξή μας ε, στο χώρο Σέγγεν. Αλλιώ θα πρέπει να προσφύγουμε στο δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να δούμε ποιο έχει δίκιο. Αλλά η παράταση αυτή τη αβεβαιότητα δίνει και μια αρνητική εικόνα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ούτε καν του ε, τους απασχολεί η κυκλοφορία ή ούτε σκέφτονται να ταξιδέψουν αλλά βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας φέρεται σαν να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις περασμένες εβδομάδες ανέφερε ότι η Βουλγαρία είναι καλύτερα προετοιμασμένη από ότι η Ρουμανία, να μπει η Βουλγαρία και η Ρουμανία όχι. Θέλω την άποψή σας. Ρουμανία-Βουλγαρία. Μπήκαν το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρηθήκαμε ένα ζευγάρι. και παντού και στις μεταρρυθμίσεις και στα κριτήρια για το Σέγγεν ήμασταν ε, μαζί στην αντιμετώπιση. Τώρα θέλετε να μας χωρίσετε, είναι άδικο αυτό. Θα πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και να ενταχθούμε ταυτόχρονα στο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ραντέμοφ, τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βασίζεται στην ενότητα και την αλληλεγγύη μας. Σε ό,τι αφορά όμως τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, βλέπουμε εδώ έλλειψη αλληλεγγύης, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ιδίως αυτές χώρες τεχνικά είναι έτοιμες να ενταχθούν ε, στο χώρο Σέγγεν. Αλλά πόρο απέχει μάλλον η ενταξή τους. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και απαράδεκτο να μην αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχουν ε, κάνει τα δύο κράτη αυτά. Έχει αποδείξει η Βουλγαρία ότι αξίζει. Έχει πολύ καλά στοιχεία στη μεταναστευτική πολιτική και φυλάσει τα εξωτερικά μας σύνορα πολύ καλά, όπως είπε ένας ομιλητής προηγουμένως, ο κ. Καρέρα. Ε, το Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει την απόφαση να ενταχθούν οι δύο χώρες, Ρουμανία και Βουλγαρία, στην, ε, ε, στο χώρο Σέγγεν. Εμείς προστατεύουμε τα εξωτερικά σύνορα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούμε στο Σέγγεν. Μάλιστα. Τώρα Έχουμε μπει στην ώρα που είχαμε προβλέψει για το δεύτερο πάνελ. Παρακαλώ, έχετε από δύο λεπτά έκαστος για να απαντήσετε στι ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Ο Dr. Καρέρα πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας που εκτιμώ ιδιαίτερως. Πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου και τον μηχανισμό αξιολόγηση ΕΝΓΕΝ. Δεν τα θέτουμε δυσβευτικά. Λέμε ότι στη νέα πρόταση τη Επιτροπή η αξιολόγηση κινδύνου είναι ένα πολύ χρήσιμο τρόπο να έχουμε μία εκτίμηση τη κατάσταση μαζί με τι γειτονικέ χώρε και αυτό είναι θετικό ε, να συμμετέχουν και οι γειτονικέ χώρε μαζί με τα κρατημέλη σε αυτή την αξιολόγηση κινδύνου. Όμω και πάλι στα χέρια των κρατών μελών βρίσκεται αυτή η αξιολόγηση κινδύνου. Των κρατών μελών που επανεισάγουν του ε, ε, ελέγχους. Γι' αυτό και δεν ξέραμε ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό είχαμε αυτό το μηχανισμό αξιολόγησης με βάση ε, έκτακτες επισκέψεις και προτείνουμε αυτό να γίνεται συστηματικά στους ε, συνοριακούς ελέγχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και αν αξιοποιούνται αναλογικά ε, με βάση την ε, διασφάλιση της ασφάλειας στην Σέγγεν. Τώρα, υπάρχει και μια σειρά θετικών ε, στοιχείων με αυτή την ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των άρθρων 25 και 29 που ξέρετε ότι η Επιτροπή χαιρετίζει την ε, ιδέα επίλυσης ή εξομάλυνσης της ε, σημερινής κατάστασης, όμως υπάρχουν και κίνδυνοι σε ό,τι αφορά το μήνυμα που αποστέλει για κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι αυτή τη στιγμή παράνομο. Είπαμε και ότι δεν υπάρχουν πλέον χρονικά περιθώρια για αυτά τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά τους συνεργούς ελέγχους. Για τους υπουργούς εσωτερικών και τι θα γίνει στο μέλλον. Εμείς λέμε ότι όσο περισσότερα τέτοια επιμένουν στην επανεσαγωγή των εσωτερικών ελέγχων, τόσο περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε για να γίνεται αξιολόγηση και να περιορίζεται και το περιθώριο λιγμών τους. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν ότι ξέρουν, να, να φροντίσουν να ξέρουν τις επιπτώσεις των πράξεών τους. Έχει παρέλθει πλέον η ε, κρίση με την έννοια και των δευτερογενών μετακινήσεων και πρέπει να επικεντρωθούμε στην σωστή εφαρμογή του κοινού συστήματος ασύλου, να εξετάσουμε τον μηχανισμό κατανομής και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη συμμορφούνται με τους υφιστάμενους κανόνες, αλλά να ασχοληθούν και με την ε, διαμόρφωση ενός νέου συστήματος. Και αυτό είναι που κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει πέραν της λογικής του συστήματος του Δουβλίνου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουάιατζο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και που στηρίζετε την ένταξη της χώρας μου στο χώρο Σέγγεν και έτσι επιβεβαιώνεται και για άλλη μια φορά η στήριξη του Κοινοβουλίου στην προσπάθειά μας αυτή. Θα ήθελα να αναφερθώ στα εξή. Επί της αρχής αρχικά, γιατί αυτό εγγράφεται και στις συνθήκες, έχουμε εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις, έχουμε κάθε δικαίωμα να συμμετέχουμε στη, στο χώρο Σέγγεν. Δεύτερον, είναι ζήτημα ενίσχυσης του χώρου Σέγγεν. Και είπαμε όλοι ότι ότι η τη ενώση από κοινού λοιπόν πρέπει να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τον χώρο Σέγγεν. Πρέπει να επιτρέψουμε στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία να ενταχθούν. Και τρίτον, και από πρακτικής άποψη, ήδη εμείς παρέχουμε ασφάλεια. Είτε ε, ήδη ε, ενεργούμε ως de facto μέλη της ΕΝΓΕΝ και είναι σημαντική η συνεισφορά μας. Για να απαντήσω τώρα συγκεκριμένα σε ένα ερώτημα που μου απίφθινε ο κύριος Κοέλιο για τα θετικά σημάδια. Εμείς ε, ως αξιωματούχοι της κυβέρνησης και διπλωμάτες πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πάντα πρέπει να βλέπουμε το φως στο τούνελ να αναζητούμε τα θετικά σημάδια και αυτό κάνουμε συνεχώς. Συνομιλούμε με εκπροσώπους όλων των κρατών μελών και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ ε, καλή παρουσία και θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες, να, θα αναδεικνύουμε συνεχώς ε, τη συμβολή μας ε, στην ασφάλεια στο χώρο Σέγγεν και συμβάλλουμε και στην αναθεώρηση και ενίσχυση του χώρου Σέγγεν. Ελπίζουμε ότι και αυτό θα είναι ένα θετικό σημάδι για την ένταξή μας στο μέλλον. Ευχαριστώ. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ε, που σας βλέπω. Ε, ποιος θα, απαντήσει τώρα, ο κύριος Γκάρκοφ. Δύο-τρία λεπτά να πατήσετε μόνο ή να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Now move to the second session. Okay, we'll with Okay, then we're moving to the second Α, προχωρούμε στο δεύτερο πάνελ από ό,τι κατάλαβα, στη δεύτερη ενότητα. Μάλιστα. Ε, αποτίμηση της λειτουργίας του χώρου Σέγγεν. Σας ευχαριστούμε που μας ήρθατε το πρώτο πάνελ. Γεια σας. Λοιπόν, αρχίζει η δεύτερη ενότητα. Έχουμε τον κύριο Σιμό Μοχτού, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, τον κύριο Μίκο Σίμολα από το ε, Υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Φιλανδίας και τον κύριο Φαμπρίς Λεζερή, εκτελεστικό διευθυντή του Frontex και του Ευρωπαϊκού ε, Σώματος Σύνοροφυλακής και Ακτοφυλακής. Yes. As we said, we're moving now to the uh, second part of this hearing. Όπως είπαμε λοιπόν, βρισκόμαστε στη δεύτερη ενότητα της ακρόασης. Καλωσορίζω στο Προεδρείο τον κύριο Σίμω Μόγδου τον κύριο Φαμπρίς Λεζερή. Καλώς για άλλη μια φορά στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Και το Σύμβουλο Μίκο Σίμολα από το Υπουργείο Εσωτερικών και ο συνιστής Φινλανδίας. Στόχος της παρούσης ενότητας είναι να εξετάσουμε την κατάσταση του Σέγγεν, ιδιαίτερα ποια είναι τα ευρήματα ε, της εφαρμογής του τροποποιημένου μηχανισμού αξιολόγησης Σέγγεν και του κανονισμού, της εφαρμογής του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θα αρχίσουμε από τα γενικά ευρήματα που θα μας παρουσιάσει ο κύριος Μοχτουρ. Άρα θα έχετε το λόγο τώρα για 10 λεπτά και στη συνέχεια οι υπόλοιποι ομιλητές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω το μηχανισμό ε, της αξιολόγησης του Σέγγεν, να δούμε τι ευρήματα έχουν προκύψει. Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι το Σέγγεν, ο χώρος αυτός είναι σαφέστατα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα και ο Επίτροπος θα σας μιλήσει για τα οράματά του για το μέλλον αλλά είναι και ένας τομέας που έχει τεράστιες προκλήσεις αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια και προσπαθούμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση και να επιτρέψουμε σε μια κανονικότητα και μια ομαλότητα. Προαπαιτούμενο γι' αυτό είναι εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ευρωπαίων πολιτών. Για ποιο λόγο το λέω αυτά. Γιατί ε, το σημαντικότερο εργαλείο ε, είναι αυτός ο μηχανισμός αξιολόγησης για να επανέλθει αυτή η εμπιστοσύνη, να και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ε, το success story αυτού του μηχανισμού και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός, ο νέος για την αξιολόγηση του Σέγγεν είναι σε λειτουργία για τρία χρόνια τώρα και αυτό μας δίνει αρκετές πληροφορίες ε, για να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα για το τι λειτουργεί καλά, τι δεν λειτουργεί καλά να σας δώσω μερικά στοιχεία και πρακτικά επιτεύγματα. Σε αυτή την τριετία τώρα έχουμε κάνει 85 επισκέψεις αξιολόγησης και εγκρίνει 85 εκθέσεις αξιολόγησης. Κάθε αποστολή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ε, έχουμε εκπροσώπους από 8 κράτη-μέλη, 2 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλο και περισσότερο παρατηρητές από τους εξωτερικούς περιφερειακούς οργανισμούς, όχι μόνο το Frontex, αλλά και τους άλλους που έχουν ρόλο να διαδραματίζουν. Τι κάνουμε εκεί στο μηχανισμό αυτό. Υπάρχει ένας αριθμός κρατών μελών που αξιολογούνται σε έξι διαφορετικούς τομείς πολιτικής ετησίω. Αυτό αρχίζει από τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, κοινή πολιτική θεώρηση, διαβατηρίων, σύστημα ενημέρωση, σέγγεν, επιστροφές, αστυνομική συνεργασία, προστασία δεδομένων. Κάτι άλλο που έχουμε, εκτός από τις ε, ε, ε, ανακοινωθήσεις ε, ε, επισκέψεις έχουμε και έκτακτες ευνηδιαστικές για να δούμε πώς εφαρμόζεται επιτόπου στα κράτη-μέλη το κεκτημένο του Σέγγεν. Ένας από τους στόχους λοιπόν ε, του μηχανισμού αξιολόγησης είναι επίσης να εξακριβώνει ότι υπάρχουν απαραίτητες προϋποθέσεις για να πληρείται ε, το ε, κοινοτικό κεκτημένο για τις χώρες που θέλουν να μπουν στο Σέγγεν και να καταργήσουν τους συνοριακούς ελέγχους. Εδώ συνδέεται αυτό με την προηγούμενη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και καιρό θεωρεί ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία πληρούν τις προϋποθέσεις. Και πέρσι και πρόπεση έχουμε εργαστεί με την Κροατία από το 2016 και το 2017 κάνουμε επισκέψεις και ελπίζω αυτό να οδηγήσει σε ένα προσεχές μέλλον σε θετικές συστάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα είναι έτοιμη και η Κροατία να ενταχθεί βεβαίως να στο Συμβούλιο να λάβει την απόφαση αυτή. Την τελευταία λοιπόν τριετία νομίζω καταφέραμε να επιδείχουμε σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της ποιότητας και της ομοιομορφίας ε, των αξιολογήσεων. Γιατί οι εκθέσεις μας είναι καλύτερες ποιότητας, πιο συνεκτικές, έχουμε ε, μια διαδικασία παρακολούθησης ε, πιο διαρθρωμένη. Ε, και τώρα και κατά τη διάρκεια των επισκέψεων είναι ένα καινούργιο θέμα αυτό που μας απασχολεί ε, να έχουμε συνδυασμένη αποστολή για την αξιολόγηση των εξωτερικών συνόρων. Όπως σας είπα, όλο και περισσότερο συμμετέχουν οι περιφερειακοί οργανισμοί, ε, Europol, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Συνοροφυλακή και Ακτοφυλακή. Και επίσης πολύ καλή δουλειά γίνεται και στην κατάρτιση και στις υπόλοιπε ε, επισκέψεις για το πώς κάνουμε την αξιολόγηση, πώς γράφουμε την έκθεση. Ε, για το θέμα των ευάλωτων σημείων θα μιλήσει κάποιος άλλος. Ε, επόμενος ομιλητής. Είναι δύο σημαντικά στοιχεία του ποιοτικού ελέγχου αυτά, δηλαδή του check-up που κάνουμε, το ελέγχου υγείας του συστήματος Σέγγεν και μάλιστα πολλές φορές είναι διόψη του ιδίου νομίσματος. Ο Φαμπρίς ε, από τη Frontex και εγώ συνεργαζόμαστε πολύ έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαλειτουργικότητα, σωστή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο εργαλείων και οργανισμός και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζονται ανα πάσα στιγμή πολύ στενά για να αξιοποιούμε και να εκμεταλλευόμαστε όσο δίνεται ε, τις συνέργειες. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Ποια είναι τα ευρήματα που επανέρχονται, που είναι συχνά ξανά και ξανά και ποιες είναι οι προκλήσεις, τα προβλήματα που έχουμε για τα κράτη-μέλη. Να δούμε στους διάφορους τομείς πολιτικής. Ας πούμε, στη φύλαξη ή διαχείριση των εξωτερικών σύνορων. Έχουμε τριών ειδών σύνορα. Χερσαία, θαλάσσια και ε, στον αέρα τι διαπιστώνουμε, ότι στα κράτη-μέλη δεν υπάρχει πάντα μια κοινή προσέγγιση, ούτε ολοκληρωμένη αντίληψη για τη διαχείριση των συνόρων. Καμιά φορά βλέπουμε προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών και αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Καμιά φορά υπάρχει και υποστελέχωση ε, στην διαχείριση των συνόρων ή έλλειψη πόρων ή όταν έχουν προσωπικό δεν είναι σωστά καταρτισμένο και δεν έχει σωστά προσόντα και δεξιότητες. Και η προσέγγιση ε, έχει να κάνει περισσότερο με την ανάλυση του κινδύνου που χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι. Όταν γίνεται λόγος για τους συνοριακούς ελέγχους, το πρόβλημα που συχνά εντοπίζουμε και είναι οι συνθήκες εισόδου οι αρχικές συνθήκες μάλλον για τον έλεγχο πολιτών τρίτων χωρών. Δεν αξιοποιούνται πλήρως πάντα οι βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες και το είδαμε αυτό με την ταυτοποίηση ε, λεγόμενων ξένων μαχητών, τρομοκρατών. Είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Στην αστυνομική συνεργασία πολύ συχνά βλέπουμε να υπάρχουν ακόμα κενά σε σχέση με την ίδρυση ε, Ενό Εθνικού Κέντρου Ανάλυσης Κινδύνου με διασυνοριακή συνεργασία. Χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση και περισσότερη στελέχωση σε μια μονοαπευθυντική θηρίδα για την αστυνομική συνεργασία. Κάτι άλλο που ακούσαμε και προηγουμένως είναι η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε ε, τράπεζες δεδομένων και ένα κοινό σύστημα διαχείρισης. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν περισσότερο και να ε, ε, κάνουν κοινέ αστυνομικές Επιχειρήσει κοινού ελέγχου. Στο SIS το μεγαλύτερο πρόβλημα και δυναμία που έχουμε εντοπίσει στις αξιολογήσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν πρόσβαση ε, ε, οι τελικοί χρήστες, πώς τους παρουσιάζεται στους αστυνομικούς, στους συνοριοφύλακες. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούν και δεν υπάρχουν μέτρα ε, συνέχεια στην εσωτερική χρήση Δηλαδή δεν χρησιμοποιούν πάρα πολύ σε εθνικό επίπεδο τις δυνατότητες που έχει το SIS. Υπάρχουν δυσκολίες ε, στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση των τελικών χρηστών. Άλλο θέμα, η πολιτική των θεωρήσεων διαβατηρίων. Να σας πω πρώτα τα καλά νέα. Ε, το βασικό που μας ενδιαφέρει και που ελέγξαμε, ελέγχουμε ε, τις αιτήσει ε, ε διαβατήριων γενικά είναι καλή αυτή, είναι ικανοποιητική. Ο τρόπος δηλαδή που γίνεται ο έλεγχο των αιτήσεων. Λίγα ήταν τα προβλήματα, οι αδυναμίε. Αυτό όμως που ε, διαπιστώνουμε πολλές φορές ως προβληματικό είναι ότι καμιά φορά τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικό τρόπο και διαφορετική κουλτούρα για τις θεωρήσει και με τον τρόπο που δίνουν βίζες. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε αγοραπολισία θεωρήσεων τώρα και πολλές φορές αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με έλλειψη προσωπικού. Ε, στο θέμα των επιστροφών το έχουμε συζητήσει, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γενικά δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τις επιστροφές και επίσης βλέπουμε ε, κάποια προβλήματα να επαρέχονται ξανά και ξανά. Δηλαδή, συστηματική έκδοση αποφάσεων επιστροφών για παράνομα διαμένοντες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ από τα κράτη-μέλη. Όπως και η απαγόρευση εισόδου. Οι κανόνες για την κράτηση, την προαναχωρησιακή, αλλάζουν και διαφέρουν πάρα πολύ από χώρα σε χώρα και επίση ε, υπάρχουν διάφορα κράτη-μέλη που δεν λαμβάνουν αρπακή μέτρα για την εκτέλεση και την επιβολή των δικαστικών αποφάσεων. Του χρόνου νομίζω θα χρειαστεί να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό ε, και στις ε, αξιολογήσεις του Σέγγερ για να προσπαθήσουμε να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Στην προστασία των δεδομένων, επίσης ένας κλάδος που σας απασχολεί πολύ στενά, ε, βλέπουμε συχνά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ε, έλλειψη ανεξαρτησίας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν υπάρχουν και ε, στοιχεία και πραγματογνωμοσύνη πολλές φορές στις αρμόδιες αρχές. Σε συστήματα VIS και SIS δεν ενημερώνονται καιρός οι ενδιαφερόμενοι για τα δικαιώματα που έχουν ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε εμείς τουλάχιστον. Είναι ο χρόνος που μας παίρνει η διαδικασία για την αξιολόγηση. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος και πλέον μετά την επίσκεψη για να καταθέσει σχέδιο δράσης η χώρα την οποία είχαμε επισκεφθεί. Ε, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία έχουν να κάνουν με τις απαιτήσει του κανονισμού. Θα το ξαναδούμε με το νέο κανονισμό, τι γίνεται με αυτές τις διαδικασίες, μήπως μπορούμε να τις απλουστεύσουμε, να τις συντομεύσουμε. Προς το παρόν προσπαθούμε να βρούμε εσωτερικές λύσεις για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Και τέλος, γιατί ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο, θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα από την πλευρά τους για να βελτιώσουν το μηχανισμό. Υπάρχουν κράτη-μέλη ε, τα οποία παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τις αξιολογήσεις και τις συστάσεις και κάνουν ό,τι μπορούν για να το αντιμετωπίσουν αυτό πολύ γρήγορα σε πραγματικό χρόνο ε, και να τα διορθώσουν άλλα κράτη-μέλη είναι κάπως πιο επιπόλαια και αργούν να υποβάλουν σχέδια δράσης ε, ή μας δίνουν σχέδια δράσης που είναι πολύ αφηρημένα, πολύ απότερα και πολύ θολά. Για μένα αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος αλλά και για τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα κράτη. Και να τελειώσω λέγοντας το εξής. Ο χώρος Σέγγεν μπορεί να είναι ε, ισχυρό, αλλά είναι ισχυρό όσο ο πιο αδύναμος κρίκο. Και είναι στο συλλογικό μα συμφέρον κάθε χώρα να ε, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιώνει το κεκτημένο. Και ο μηχανισμό αξιολόγηση έγκαινα έχει εδώ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μόρτζιου. Συνεχίζουμε. Ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σέγγεν είναι κοινή ευθύνη ανάμεσα στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Σιμόλα θα μας ενημερώσει για τη λειτουργία του μηχανισμού. Παρακαλώ, κύριε Σιμόλα, έχετε το λόγο. Έχετε 10 λεφτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, καταρχάς με μεγάλη χαρά χρησιμοποιώ αυτήν την ευκαιρία για να παρουσιάσω την άποψη των κρατών μελών για τον μηχανισμό αξιολόγηση και παρακολούθησης του Σέγγεν. Και είμαι πεπισμένο ότι η συμμετοχή μου σε διάφορες αποστολές αξιολόγησης του Σέγγεν ως βασικός εμπειρογνώμονας από την πλευρά των κατών μελών, η εμπειρία που έχω ως εκπαιδευτή στη Frontex οργανώνοντας μαθήματα για τους αξιολογητές του Σέγγεν, καθώς και η δουλειά που έχω κάνει στο παρελθόν στην Επιτροπή Σέγγεν και εν συνεχεία στην Ομάδα Εργασίας Αξιολόγησης του Σέγγεν στο Συμβούλιο, ε, είναι μια καλή βάση για να παρουσιάσω αυτή την αξιολόγηση. Θα αναφέρω κάποια γενικά πορίσματα ε, που έχουν προκύψει από επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να πω από την αρχή ότι παρουσιάζω αυτά τα θέματα με βάση τη δική μου εμπειρία που σας περιέψα πιο πριν. Λόγω αυτού του πλαισίο από το οποίο προέρχομαι, θα εστιάσω ε, στα διδάγματα που έχουμε συγκεντρώσει σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι παρότι η έλεγχη στα εξωτερικά σύνορα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία, παράλληλα είναι μόνο ένα τμήμα ολόκληρου του συστήματο Σέγγεν. Ο αποτελεσματικό έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα είναι ακρογωνιαίο λήθο προφανώ. Αλλά όμω όλη η αλυσίδα θα πρέπει να λειτουργεί καλά. Φερρυπίν το να εντοπίζουμε όλους εκείνους που διέσαλεχο στα εξωτερικά σύνορα είναι ακρογωνιαίος λίθος προφανώς. Αλλά όμως όλη η αλυσίδα θα πρέπει να λειτουργεί καλά. Φερρυπίν. Το να εντοπίζουμε όλους εκείνους που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα παράνομα. Αυτό όμως δεν αρκεί για να λειτουργεί το σύστημα, εάν το σύστημα επιστροφών δεν λειτουργεί καλά. Ε, θα ξεκινήσω παρουσιάζοντας την εμπειρία μου και τα πορίσματα ε, με βάση τα όσα λειτουργούν καλά στο σύστημα. Καταρχά, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τη Κομισιόν πάει καλά και έχει βελτιωθεί και βελτιώνεται σύν το χρόνο. Ε, ο συνολικό συντονισμό είναι πολύ καλά οργανωμένο. Θα ήθελα να αναφέρω επίση, επευκαιρία, ότι ο μηχανισμό αξιολόγηση των ευάλωτων σημείων ε, δημιουργήθηκε με βάση τον κανονισμό ε, για την Ευρωπαϊκή Συνοριαφυλακή και Ακτοφυλακή και ένα σημαντικό συμπροματικό στοιχείο ολόκληρου του μηχανισμού αξιολόγηση του Σέγγεν. Θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Δεύτερον, το σύστημα κατάρτισης και εκπαίδευση είναι ένα καλό στοιχείο. Ε, τα κράτη-μέλη οργανώνουν τα μαθήματα κατάρτισης των αξιολογητών του Σέγγεν ε, με τη βοήθεια της Κομισιόν και το Frontex και αυτό είναι ένα πολύτιμο πακέτο που συνεισφέρει στην υψηλή ποιότητα και στον επαγγελματισμό των αξιολογητών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο εκείνα τα άτομα τα οποία πέρασαν επιτυχώς το μάθημα μπορούν να επιλεγούν από την Επιτροπή για να συμμετέχουν σε ομάδες αξιολόγησης του Σέγγεν. Θα πάω τώρα στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου. Τι θα πρέπει να βελτιωθεί στο τρέχον σύστημα. Ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι η όλη διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αργή και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε όλοι μας πόσο γοργά αλλάζει η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα. Στο, με το τρέχον σύστημα, επί παραδείγματι, χρειάζεται ένας χρόνος και. Ε, αυτή τη στιγμή γίνει η επίσκεψη αξιολόγησης για να συζητηθεί η έκθεση ε, αξιολόγηση στην Επιτροπή Σέγγιν. Και οι συστάσεις ε, προς το αξιολογούμενο κράτος μέλος μπορούν να δοθούν από το Συμβούλιο μόνο όταν εγκριθεί η έκθεση. Επομένως, έχουμε μακρές καθυστερήσεις που είναι τέτοιου τύπου, που δεν είναι καλό για τον κοινό χώρο Σέγγιν. Και βεβαίως κάτι τέτοιο δεν αυξάνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών Σέγγιν. Γιατί το σύστημα είναι τόσο αργό. Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι γι' αυτό. Οι πόροι του αρμόδιου τμήματος ε, της Κομισιόν, του καθήλυνα αρμόδιου τμήματος Κομισιόν είναι, περιορισ... είναι περιορισμένη. Και η διαδικασία εσωτερικής διαφούλευσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ολοκληρωθεί η έκθεση κρατάει πάρα πολύ. Οι περιορισμένοι πόροι της Κομισιόν επίσης έχουν αρνητική επίπτωση στη συνέχεια που θα δοθεί στην παρακολούθηση για να δούμε το πώς δηλαδή, τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τις συστάσεις ε, με βάση τα πορίσματα. Μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε αυτό το follow-up, στη συνέχεια δηλαδή, ε, μετά την αξιολόγηση. Γιατί ε, περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό γίνεται αυτό το, υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, για να βελτιωθεί το επίπεδο και η ποιότητα των ε, συνοριακών της επισκέψης. Αυτό οφείλεται στις τρέχουσες τεχνικές και νομοθετικές τροχοπέδες που υπάρχουν και που αντιμετωπίζουν ορισμένε υπηρεσίε, όπω το Ιουλίζα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιτόπιε ομάδε δεν έχουν πρόσβαση σε, όλη τη, σε όλε τι ε, απαραίτητε πληροφορίε που θα χρειαζόντουσαν για να αξιολογήσουν τη λειτουργία στα κατά τη διάρκεια των αποστολών αξιολόγηση του Σέγγεν, στα εξωτερικά σύνορα πάντα, έτσι. Και θα μιλήσω για αυτά τα πορίσματα με γενικό τρόπο, γιατί δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειε. Ε, μιλάμε για πορίσματα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ξεκινάω πάλι από τα θετικά στοιχεία, από τα θετικά πορίσματα οι σύνοριοφύλακοι να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τα, τις ικανότητές τους ε, και να βρίσκουν νέες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Εν συνεχεία, θέλω να αναφέρω κάποια προβλήματα όπου χρειάζεται βελτίωση σε πολλά κράτη-μέλη. Η γνώση των κανόνων σε της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου και δεν έχουν αρκετά ε, αρκετέ ικανότητε οι συνολιοφύλακε για να εντοπίσουν τα πλαστογραφημένα έγγραφα. Το πιο όμω ανησυχητικό πόρισμα είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκεί ε, πόροι και επαρκή υποδομή στα σύνορα, στα σημεία να εγγυηθούν μέσα στα πλαίσια αυτών των περιορισμένων πόρων και υποδομών τη σωστή εφαρμογή της νέας ενωσιακής νομοθεσίας, όπως την τον υποχρεωτικό έλεγχο ε, βάσεων δεδομένων ε, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμογή του συστήματος ε, εισόδου-εξόδου και, μέχρι το 2020 και εφαρμογή του συστήματος δομές στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Γιατί αυτά τα αρνητικά πορίσματα ε, τα βρίσκουμε πολύ συχνά ε, σε αποστολές αξιολόγησης. Για ποιο λόγο. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι σε κάποια κράτη-μέλη ε, το, σύστημα, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων είναι κατακαιρματισμένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου ε, δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι σε εθνικό επίπεδο, όπου η εποπτεία και η ε, έλεγχη ε, για τον έλεγχο των συνόρων υπό την αρμοδιότητα του αρμόδιου Υπουργείου δεν υπάρχει, τότε δεν είναι σωστό. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν οι συνοριακοί έλεγχοι με βάση τη ε, σωστή κατάρτιση των συνοριοφυλάκων. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Μερικές φορές λείπει και η κατάρτιση για τους συνοριοφύλακες και αυτό οδηγεί σε κενά και σε διαρθωτικές αδυναμίες. Για να επιληθούν αυτά τα θέματα και να βελτιωθεί η κατάσταση πρέπει να συζητηθούν αυτά τα σοβαρά πορίσματα πιο ανοιχτά. Παραδοχή ότι υπάρχουν αυτά τα κενά ε, με, και να χρησιμοποιήσουμε σωστά, σωστούς και καλούς ε, αξιολογητές, επαγγελματίες για θέματα Σέγγεν. Ε, το να βρεθούν λύσει και να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα ε, δεν θα πρέπει να τα αφήσω. Σειράσω τώρα τρία σημεία για την ενίσχυση τη αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αξιολόγηση του Σέγγεν. Καταρχά, οι διαδικασίε Δηλαδή, η υιοθέτηση των ε, εκθέσεων και οι συστάσεις ε, εντοπίζουν ε, κενά και προβλήματα. Και ενδεχομένω, εάν δεν υπάρξει διορθωτικό μέτρο, να υπάρχει και διαδικασία επιπαραβάσης του κράτου. Ε, για τον, την αξιολόγηση του Σέγγεν, θα πρέπει να μας βοηθάει με έναν ευρύ. Στον επόμενο προσκεκλημένο μας που είναι πάντα ευπρόσδεκτο ο κύριος Λετζέρη, εκτελεστικός διευθυντής ε, της Ευρωπαϊκής Φορέα και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, θα προσπαθήσω να σας ε, ενημερώσω για την ε, τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νέας εντολής της Frontex υπό τη μορφή της νέας ε, ακτοφυλακής και συνεργοφυλακή και θέλω να σας επισημάνω και τη διασύνδεση με το χώρο Σένγκεν και την εφαρμογή της νέας εντολής. Τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές είναι σημαντικά και με βρίσκουν σύμφωνο σε ό,τι θα τα παρουσιάσω και εγώ στη συνέχεια, ιδίω ό,τι αφορά την αξιολόγηση για τον ευάλωτο χαρακτήρα. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι η υλοποίηση της ε, νέας εντολής και η τελευταία αυτή πτυχή που αφορά την αξιολόγηση του τροτού χαρακτήρα, η ανάπτυξη των ε, ε τετραμένων αξιωματούχων προς τα κράτη-μέλη είναι στρατηγική εξέλιξη η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά υπάρχει μία δυναμική εξέλιξη και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, εντολής και ο σχετικός κανονισμός δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή για Συνοριοφυλακή. Αυτό σημαίνει ότι από κοινού, ο οργανισμός δηλαδή, από κοινού με τις εθνικές αρχές ε, αρμόδιες για ζητήματα της ακτοφυλακής και είμαστε και οι δύο από κοινού. Πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε προς αυτό τη στρατηγική μας, τις προτεραιότητές μας, σταδιακά όλα αυτά, τη μέθοδο λειτουργίας μας και θα πρέπει να, γίνει, να γίνεται αυτή η συζήτηση, αυτός ο διάλογος ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση για τον τροτό χαρακτήρα, είναι ένα εγχείρημα ε, που συμπληρώνει τον μηχανισμό αξιολόγησης Σέγγεν, το λεγόμενο Σαβάλ, από με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Home, έχουμε ε, καθιερώσει ορισμένε ε, διόδου ανταλλαγή πληροφοριών για να αποφεύγουμε τι αλληλεπικαλύψει, ορισμένα ζητήματα και σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων. Υπάρχει στενή συνεργασία και για την κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο οργανισμός συνήθως ε, συμμετέχει στον μηχανισμό αξιολόγησης Σέγγεν και ε, υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία των αποστολών. Προτείνουμε επίσης ε, και επισκέψεις και πού πρέπει να γίνονται, ιδίως ό,τι αφορά τις μη προβλεπόμενες. Τώρα για τον νέο μηχανισμό που θεσπίστηκε πριν από 1,5 χρόνο. Είχαμε τον πρώτο ετήσιο κύκλο το 2017 σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του χαρακτήρα. Ο οργανισμός αξιολόγησε 29 κράτη-μέλη, δηλαδή ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες. Και το συμπέρασμα είναι, και εγώ προσωπικά εξέδωσα 37 συστάσεις προς 27 κράτη-μέλη. Έχουμε διάφορες κατηγορίες συστάσεων. Θα ήθελα εγώ να σταθώ στις βασικές. Σε πολλά κράτη-μέλη είδαμε ότι η απλή συνοριακή έλεγχη στα σημεία διέλευσης δεν συμμορφούνται πάντα με τις βασικές ε, προϋποθέσεις ε, που θεσπίζει ο κώδικας Σέγγεν. Η πρόσβαση στο SIS, ε, στο VIS, δεν συνάδουν πάντα με το νομικό μας πλαίσιο. Και αυτό γύρει μια σειρά ζητημάτων σε ό,τι αφορά την χρηστή διαχείριση και της μετανάστευσης και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ελεύθερη κυκλοφορία. Χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας και χώρος ε, ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μια άλλη κατηγορία αφορά τις περιορισμένες ε, δυνατότητες για την υποδοχή τεράστιων κυμάτων μεταναστών και προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα. Είπαμε λοιπόν ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν υπάρξει επενδύσεις σε αυτό το θέμα και έτσι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να υποδεχθούν ε, σημαντικά αλλά θεωρητικά διαχειρίσιμα κύματα μεταναστών. Ένα άλλο έβριμα, σημαντικά αλλά θεωρητικά διαχειρίσιμα κύματα μεταναστών ένα άλλο έβριμα σύνορα, αλλά και τη δυνατότητά μας να διαχειριζόμαστε ζητήματα ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα. Το πίση, αλλά εξίσου σημαντική, αφορά την ανεπαρκή διαχείριση ε, πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το ανέφερα για κάθε κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη ε, συντονισμού και κατά πιθανότητα και έλλειψη κατευθύνσεων ή καθοδήγηση σε εθνικό επίπεδο. Αυτό μας έκανε εντύπωση. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους από τα κράτη-μέλη προ το εγχείρημα αυτό, προ την αξιολόγηση του ροτού χαρακτήρα. Δεύτερον, το πεδίο και η μεθοδολογία ε, θα πρέπει να διευρυνθούν. Θα θυμάστε ότι αυτό το εργαλείο είναι κάτι το οποίο υιοθετήθηκε από το Διοικητικό σε ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ασφαλείας και για να αξιολογήσουμε ε, τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές ε, διαχειρίζονται τις ε, απειλές της τρομοκρατίας και των παράνομων οργανών. Είναι κάτι το ανησυχητικό, γιατί βλέπουμε ότι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στη Σένγκεν δεν είναι μόνο, και το, η πρόκληση μάλλον, δεν είναι η μετανάστευση. Είναι και το θέμα της ασφάλειας. Τα εξωτερικά σύνορα μπορούν να ενεργήσουν ως ε, κάποιο... Τα κράτη-μέλη θα πρέπει πιο γρήγορα να ανταποκρίνονται και να αντιδρούν στις, ε, στα ευρήματά μας. Παρακολουθούμε τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις μας, αλλά κάποιες φορές είναι μακροχρόνια η διαδικασία και αυτό μας δείχνει ότι κάποια απόκριση καταφέραμε να ενισχύσουμε τις δραστηριότητε μας. Σε βασικές μας επιχειρήσεις είναι η Ποσειδόν στην Ελλάδα, η Θέμη στην Ιταλία, η Ίνταλο στην Ισπανία, που είναι μόνιμη επιχείρηση αυτή τη στιγμή λόγω της αύξηση των μεταναστευτικών ροών από το Μαρόκο δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση ε, στην λήψη δεκτυλικών αποτυπωμάτων, ε, το screening στα hotspots, spots, στήριξη των κρατών μελών σε συγκεκριμένες δραστηριότητε ε, debriefing και πληρούμε απόλυτα και την εντολή μας σε ό,τι αφορά την ακτοφυλακή. Έχουμε την έρευνα και την αναζήτηση και διάσωση, αλλά ε, πρέπει να ενισχύσουμε και τις ε, λειτουργίες μας ε, στο πλαίσιο της ακτοφυλακής, μαζί και με τον, τον Οργανισμό Ασφάλειας στη Θάλασσα. Όλα αυτά είναι πολύ βασικά για να έχουμε αξιόπιστο μηχανισμό διαχείριση τη μετανάστευση ε, και έναν ε, ασφαλή χώρο Σέγγεν. Εδώ ο οργανισμός μας έχει εξοπλίσει την ε, εντολή, έχει ενισχύσει τη στήριξη σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση παράτυπων μεταναστών, τη συνεργασία με τρίτες χώρε και σε ό,τι αφορά τις επιστροφές. Έχουμε διοργανώσει πάνω από 340 πτήσεις επιστροφής πέρυσι, αύξηση 50% σε σχέση με το 2016 σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια. Σκεφτείτε ότι τότε είχαμε ε, μόλις 39 τέτοιε πτήσεις, έχουν δεκαπλασιαστεί λοιπόν. Τώρα, να σταθώ στη διεθνή συνεργασία, που εντάσσεται επίση ε, στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης συνόρων. Μια καλύτερη εικόνα των συνόρων και θέλουμε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση στην μια καλύτερη εικόνα των συνόρων και θέλουμε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση. Στην ευκαιρία έχουμε τώρα με το ε, περχόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη τα πορίσματα, τα ευρήματα, το ε, ε, τον εξοπλισμό και την συνολική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λετζέρη. Όπως πάντα εντυπωσιακός και εντυπωσιακή η ενημέρωση αυτή σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή ανταπόκριση του οργανισμού που παλαιότερα ήταν, λεγόταν Frontex, τώρα ακούσουμε και τον ε, αντίκτυπο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά την εντολή σας, με αυτόν τον πολλαπλασιασμό των ε, πτήσεων επιστροφών που δημιουργεί προβλήματα, δείχνει όμως ότι υπάρχει μια Ας περάσουμε λοιπόν σε έναν γύρο ερωταπαντήσεων. Κύριε Κοέλιο, να ξεκινήσουμε από εσάς. Έχουμε μακρύ κατάλογο μιλητών. Προτείνω λοιπόν να συνομεύετε για τους τρεις ομιλητές μας. Συμφωνώ με τον αναπληρωτή γενικό Σέμ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Task Force. Ε, πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμη η συνεργασία μας με πολύ καλά αποτελέσματα. Όμως, και για σας και για τον κύριο Σίμολα έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Σούμε ότι είναι εργαλείο. Έχει το SIS, ε, και το μηχανισμό αξιολόγησης. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Μας έχει φάει η κρυψίνια. Όλα, με τέτοιος μηχανισμός, όταν έχουμε τόσο, τόση χημήθεια, ε, δεν το καταλαβαίνω. Ο κύριος Σίμουλα μίλησε για μεγάλες καθυστερήσεις. Ε, συμφωνώ με αυτό που λέτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων και σωστά ερμηνεύω ότι τι περισσότερε φορές ε, το σχέδιο συστάσεων προ τα κράτη-μέλη και η έκθεση ε, ταυτόχρονα έρχονται ε, στην Επιτροπή μας. Και προς τον κύριο Λετζέρη, καταλαβαίνω ότι η πλαστογράφηση των εγγράφων είναι πρόβλημα, αλλά συμφωνείτε ότι μπορούν τώρα οι αστυνομικέ δυνάμεις μας στα σύνορα να ανοιχνεύουν τα πλαστά έγγραφα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το πρόβλημα είναι κάποια έγγραφα ε, τα οποία έχουν εξαιρετική ποιότητα πλαστογράφησης. Μπορεί να φαίνονται γνήσια, αλλά είναι πλαστά. Το ξέρω ότι δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Όλο το μέλη του πάνε. Κυρία Κραπίνη. Ευχαριστώ πολύ. Βιολόγηση δεν ε, μας χαροποιούν μόνο, αλλά μας ανησυχούν πολλές φορές. Ε, πάντως μας δώσατε συγκεκριμένα στοιχεία και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Να κάνω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Γιατί με προβλημάτισαν πολύ αυτά που είπατε. Και πώς εκτιμάτε την εξωτερική, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ε, ενώ υπάρχουν χώρες που δεν είναι ε, μέλη του Σέγγεν. Είπα του Σέγγεν. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ποιο είναι ο στόχο, η σωστή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Αλλά δεν έχουμε του κατάλληλου μηχανισμού στα χέρια μα πάντα. Επίση, είπατε και οι τρει ότι ο μηχανισμό ε, ακόμα δεν είναι ιδεώδε, κάποια κράτη-μέλη καθυστερούν, χρονοτριβούν υπάρχει καμιά κατάσταση. Επίσης μιλήσατε για τα κράτη-μέλη που δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ε, τις αξιολογήσεις. Ποια είναι τα κράτη-μέλη αυτά, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικώ. Τα κράτη που ανήκουν στο χώρο Σέγγεν, τα κράτη που περιμένουν, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Συμφωνώ με αυτό, όσα είπε ο κύριος Κοέγιο, ότι όλα αυτά Πολύ ωραία τα διαπιστώνουμε εμείς, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα να τα βγάλουμε προς τα έξω και τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος μας. Που είναι η διαφθορά ένας από τους αδύναμους κρίκους. Δεν είναι ότι δεν τα γνώρισε Σέγγεν και καλά ε, ε, το έκαναν, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι είχαν πάρει κανονική βίζα Σέγγεν. Αυτό τι σημαίνει, δεν υπάρχουν πόροι, ότι προφανώς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους για να γίνεται σωστά αυτή η αξιολόγηση και αποτελεσματικά, αλλά ελπίζω να μην συμβαίνει το ίδιο με τις δικές σας εκθέσεις για την αξιολόγηση του μηχανισμού Σέγγεν ή μήπως συμβαίνει. Πείτε μας παρακαλώ τι συμβαίνει. Κάνουν καμιά διαφορά, βελτιώνουν τα πράγματα εκθέσεις σας. Επισημαίνετε κάποια πράγματα, τα διορθώνουν τα κράτη-μέλη. Ερώτηση δεύτερη. Και μόνο. Αλλά υπάρχουν διαφορετικές αρχές. Στη Μάλτα, ένα μικρό κράτος μέλος, πρόσφατα είχαμε μια αποστολή κράτους δικαίου και διαπί. και αυτό που λένε έπιπη που είναι ηθαγένεια, υπηκότητα. Τους ξέρετε αυτούς, εκεί συνεργάζεστε που έχω στα χέρια μου για ένα σύστημα που έχουν στήσει εκεί και πουλάνε βίζε Σέγγεν σε Λίβιους στη Μάλτα. Αυτά τα θέματα σας απασχολούν, τα ψάχνετε. It's not just... Δεν είναι μόνο η Μάλτα. Ούτε πρόκειται μόνο για τη Μάλτα. Για όλους εμάς πρόκειται. Είναι πολύ σοβαρές περιπτώσεις όταν συμβαίνουν στις χώρες μας αυτές, αναρωτιέμαι. Τα έχετε αντιμετωπίσει αυτά. Θα σας δώσω πληροφορίες πάρα πολύ σύντομα. Η κυρία Βεργιά. Merci, Monsieur le Président. Στο πρόεδρε. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι μεγαλίδα, αλλά διάφορα πράγματα ε, επιστροφών, που είναι ένα μείζον στοιχείο βέβαια των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών σήμερα. Εγώ εξακολουθώ να παραμένω ανήσυχη συνεδρίαση. Το βασικό θέμα, ε, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να πάμε στο βασικό χερσαίο σημείο διέλευση που είδαμε να γίνονται στα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Και... Ε, υπάρχουν κάποιες ώρες εχμής, ας πούμε, στην πρωτεύουσα ε, και χαλαρώνουμε τους ελέγχους. Όχι, ε, μειώθηκαν δικά κατά 80%. Ε, το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές, γιατί οι, τρομε, ε, οι τρομοκράτες τμήμα και μέλημα της αξιολόγησης, γιατί νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό ε, στα πλαίσια του δικαιώματος ασύλου και του δικαιώματος υποβολή κοινοβούλου. Έτσι δεν είναι πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Βερσιά στο επόμενο πάνελ έχουμε και τον Επίτροπο ε, Αβραμόπουλο και τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, κυρία Βεωσία. Ε, Θέλω λοιπόν, ε, πριν τελειώσει αυτό το πάνελ, να δώσω τουλάχιστον για δύο λεφτά τους ε, τωρινούς πανελίστες το λόγο για να απαντήσουν. Οπότε να το έχετε υπόψη όταν διατυπώνετε τις ερωτήσεις σας. κυρία Πίνμπερκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και το πάνελ στο σύνολό του. Είναι πολλές οι ελλείψεις λοιπόν και αδυναμίες που ε, διαπιστώσατε στο σύστημα Σέγγεν. Είναι καλό ε, τουλάχιστον να ενισχυθεί η συνεργασία στο χώρο Σέγγεν και επίση θα ήταν ακόμα καλύτερο να μπορούσαμε να καταργήσουμε όλους τους εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λειτουργήσε πολύ καλά για πολύ χρόνο. Τώρα όμως τι διαπιστώνουμε, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να έχει και μειονεκτήματα, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα πλεονεκτήματα. Λαθρεμπόριο, εγκληματικότητα, κανένας έλεγχος για το ποιος ε, εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος κυκλοφορεί στα κράτη, από το ένα κράτος στο άλλο. Γι' αυτό είναι ε, γεγονός αυτή η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει κάποια προβλήματα στο παρελθόν εάν είχαμε διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους. Όχι, θα πρέπει να είναι μόνιμοι για να καταγράφονται οι πάντες. Με τις τεχνολογίες που διαθέτουμε γίνονται όλα αυτά πιο γρήγορα από ό,τι στη δεκαετία του 90. Τα διαβατήρια πια ελέγχονται αυτόματα, συντομότεροι. Να αρχίσουμε με την αντίστροφη σειρά. Ε, μάλλον, ε, ε, ε, απαντήστε εσείς κύριε Λεζερή Για τις πτήσεις επιστροφών, ποιοι είναι οι προορισμοί, οι συνηθέστεροι και τα αεροδρόμια από το... Ξεκινώ με το ερώτημα του κύριου Κοέλιο. Νομίζω ότι ήδη η σημερινή συζήτηση είναι σημαντικό βήμα. Μας δίδεται έτσι μοιάσουμε ενιαία έναν αριθμό βασικών ε, ευρημάτων ε, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση Σέγγεν. Γιατί όντως υπάρχει, ε, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε στα κράτη-μέλη και βλέπουμε ότι εν γέννη η κατάσταση βελτιώνεται και είναι σημαντικό αυτό. Τι προποθέσει και ελπίζουμε να τι υποδεχθούμε σύντομα στη ζώνη Σέγγεν. Τώρα, κάτι το οποίο έχουμε δει αρκετά συχνά ε, στο προκλήσει και με τι γειτονικέ μα χώρε, και εργαζόμαστε όσο μπορούμε για να συνάψουμε επιχειρησιακέ συμφωνίε με κάποιου από του εταίρου μα στα Δυτικά Βαλκάνια στις επιτόπιες επισκέψεις μας. Αξιολογούμε όλους τους φορείς που ε, ενεργούν στο πλαίσιο του συστήματος. Προσοχή όμως εδώ. Ο μηχανισμός αξιολόγησης Engen εξετάζει τη δομή, την οργάνωση και τις επιχειρήσεις. Δεν είναι ε, μηχανισμός δίωξη. Εξετάζουμε και τα εσωτερικά σύνορα μεταξύ κρατών μέλων και όχι μόνο τα εξωτερικά. Και γιατί το κάνουμε αυτό γιατί με τον κατάλληλο τρόπο στις ε, απειλές προς τη δημόσια τάξη ε, και την ασφάλεια. Παράλληλα όμως, η μόνιμη είναι ε, ένα έκτακτο μέτρο, μια εξαίρεση, μέτρο τελευταίας ανάγκης και να έχουμε άλλες εναλλακτικές όπου αυτό είναι δυνατόν. Έτσι θα ήθελα να κλείσω. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Σίμολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ξεκινώ από τις ερωτήσεις του κ. Κοέλιο. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καθυστερήσεις. Είπα ότι έχουμε το νομικό μας πλαίσιο και να λάβουμε υπόψη όλα όσα έχουμε μάθει από το παρελθόν. Για να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι συμβαίνει από εδώ και πέρα, στο follow-up της ε, δομές του Συμβουλίου. Επομένως, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη και οι δύο συμπειρογνώμονε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Άσμου ξέρουμε ότι είναι ε, πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ε, ω έλεγχο έλεγχος και όλα αυτά πρέπει να επηρεάσουν την ε, κρίση. Είπε ο κύριος ε, Λεζερή ότι είναι και ένα φίλτρο στα σύνορά μας η διαχείριση των σύνορων ή μάλλον η έλεγχη στα σύνορα. Έχουν δυνατότητε βελτίωση και με την ε, βελτίωση της συνεργασίας για την καταπολέμηση του διασυνορικού εγκλήματος. Γιάνονται περισσότερο στους ε, κακοί τυπίστοι ταξιδιώτες και όχι στους καλοί τυπίστοι ταξιδιώτες. Και ως... ...του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε εξ ονόματος της Προεδρίας τον ε, Υπουργό Βαλεντίν Ράντεφ, Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας. Σας καλωσορίζω και σας θερμά στην Επιτροπή μας δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα και κάτι. Και επίση έχουμε και δώσω το λόγο στον κύριο Κοέγιο που ήταν ε, ο εισηγητής για τον κανονισμό για την αξιολόγηση του Σέγγεν και τώρα είναι ο εισηγητή για τον κανονισμό για το SIS. Ο κύριος Κοέγιο επίσης είναι και πρόεδρος της ομάδας εργασίας μας για τον έλεγχο του Σέγγεν. Παρακαλώ κύριε Κοέγιο. ξεκάθαρα. Κι όμως, να ακόμα μία παράταση ανάμεσα στην ε, Γερμανία και στην Αυστρία. Γερμανία και Αυστρία δηλαδή ζήτησαν κάτι τέτοιο τη στιγμή που δεν υπάρχουν επιχειρήματα, δεν έχουμε παράνομες διαλέψει. Είναι πολύ δύσκολο να πείσω στη δική μου χώρα την... Ε, και ελπίζω να μην... Και δεν νομίζω ότι είναι ε, το μπαλάκι στη... Ε, στο Κοινοβούλιο, αλλά στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Υπουργέ. Καταρχά θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τα μηνύματα του Κάρλος και της Τάνια. Προσωπούν και εκφράζουν την ισχυρή στήριξη του Κοινοβουλίου για το Σέγγεν. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ελεύθερη κυκλοφορία, όπως γνωρίζετε, είναι εγενές ε, χαρακτηριστικό των καιρών μας και στο μέλλον δεν μπορεί παρά να αυξηθεί με όλες τις, τις εκφάνσεις. Έχουμε όλοι συμφέρον να το ενθαρρύνουμε αυτό, αλλά και να το διαχειριστούμε. Επανειλημμένα έχει υποθεί ευθύ εξ αρχής ότι το Σέγγεν είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα και τα πιο χειροπιαστά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για να μην πω το μεγαλύτερο. Η αποσία εσωτερικών συνοριακών ελέγχων συνιστά την πεμπτουσία του πνεύματος του Σέγγεν. Πάνω από 400 εκατομμύρια πολίτες και επισκέπτες μπορούν ελεύθερα να μετακινούνται. Υπηρεσίες, αγαθά μπορούν να ρέουν απρόσκοπτα. Αλλά και πολύ περισσότερο, πέρα από όλα τα λογικά επιχειρήματα και τα οικονομικά ωφέλη, ο χώρος Σέγγεν αποτελεί σύμβολο για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στο Σέγγεν έχουν καταργηθεί τα σύνορα μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Τα ίδια ακριβώς σύνορα τα οποία στο παρελθόν οδήγησαν σε διενέξεις, σειράξεις, συγκρούσεις και πολέμους. I have lived. Ως νεαρός παρακολούθησα τις αλλαγές από τα σύνορα που υπήρχαν τότε μέχρι την κατάργηση των εσωτερικών σύνορων. Οι νεότερες γενιές το θεωρούν δεδομένο πλέον αυτό. Πιστέψτε με, δεν ήταν καθόλου προφανές αυτό πριν από τρεις δεκαετίες μόλις. Ως επίτροπος και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το λόγο αυτό είμαι απόλυτα προσιλωμένος στην διαφύλαξη και στην ενίσχυση του Σέγγεν. Και θέλω να εξασφαλίσω ότι θα συνεχίσει να μας δίνει τα ίδια ωφέλη και στο μέλλον. Το Σέγγεν έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και σε πολλές περιπτώσεις απειλές. πρωτοφανείς μεταναστευτικές προκλήσεις, τις οποίες αντιμετώπισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση επί μία διετία και πλέον. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη πίεση για το Σέγγεν και τη λειτουργία του από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Διάφορα κράτη-μέλη έχουν επαναφέρει εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους προσωρινού χαρακτήρα σε μια απόπειρα να ρυθμίσουν και να ελέγξουν κάπως την παράτυπη μετανάστευση και αντιδρώντας στις πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις. Πλην όμως η προσωρινή εσωτερική συνεργειακή έλεγχη δεν επιτρέπεται και δεν θα πρέπει να καταστούν μόνιμοι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε για να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εξασφάλιση της κυκλοφορίας από τη μία και την εγγύηση της ασφάλειας από την άλλη. Ακριβώς για να διατηρήσουμε την ισορροπία αυτή προτείναμε να τροποποιήσουμε τον συνοριακό κώδικα του Σέγγεν. Υπάρχει κάτι που είναι ξεκάθαρο τα κράτη-μέλη διατηρούν τη βασική ευθύνη ως προς το θέμα της ασφάλειας. Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, θα πρέπει να μιλήσουμε ότι η προσωρινή επαναφορά συνοριακών ελέγχων είναι ένα μέσο νόμιμο και θεμητό που έχουν στα χέρια τους τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές για την εσωτερική τους ασφάλεια, τη δημόσια τάξη σε έκτακτες περιπτώσεις. Πρόθεσή μας όμως δεν είναι η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων να καταστεί ευκολότερη, πόσο μάλλον μόνιμη. Το αντίθετο. Αυτό που εμείς προτείναμε είναι να ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω ε, τις δικονομικές ε, ασφαλιστικές δικλείδες ή τις διαδικασίες η επαναφορά των ελέγχων αυτών θα πρέπει να είναι μέτρο εσχά της καταφυγής και μόνο. το τελευταίο λόγο του έχει το Συμβούλιο και οι απόψει των άλλων κρατών μελών επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δε όντως, των κρατών που θίγονται από τέτοιου είδους αποφάσεις επαναφοράς συνοριακών ελέγχων. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ακόμα το εξή. Είναι σαφώς πολιτικό αυτό το θέμα. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο εσωτερική πολιτικής. Ποιε είναι εναλλακτικέ λύσει. Αστυνομική έλεγχη, διασυνοριακή συνεργασία. Αυτές θα πρέπει πάντα να έχουν την προτεραιότητα. Ελπίζω να βρούμε γρήγορα ένα συμβιβασμό για την πρόταση αυτή που κατά την άποψή μας συνιστά μια πολύ προσεκτική ισορροπία όλων των θεμητών μας ε, συμφερόντων. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει μετά να αρχίσουν να ισχύουν και θα μας επιτρέψουν να αποτρέψουμε τις καταχρήσεις και να βεβαιωθούμε ότι όλοι τηρούν τους κανόνες. Στα πλαίσια αυτά προσβλέπω στην ανάγνωση της έκθεσης κυρίας Φαγιών επί της ε, νομοθετικής ε, τροποποίησης που προτείνουμε. Ταυτόχρονα, όπως όλοι γνωρίζετε, η κυκλοφορία εντός των συνόρων μας απαιτεί ασφαλή εξωτερικά σύνορα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, από το 2015, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των μεταναστών που φτάνουν από την Ανατολική Οδό και την Οδό της Κεντρικής Μεσογείου έχουν μειωθεί δραστικά. Ένα βασικό στοιχείο ήταν η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Σύνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που τώρα είναι πλήρως επιχειρησιακή. Αυτή τη στιγμή ο οργανισμός αναπτύσσει ε, περίπου 1.200 σύνοριοφύλακες για να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα με επιπλέον 1.500 που προβλέπονται και είναι σε επιφυλακή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την απουσία των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη φύλαξη των εξωτερικών μας συνόρων. Επίσης, κάτι άλλο που χρειαζόμαστε είναι να αποφασίσουμε εάν θα διατηρήσουμε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως έχει ή μήπως θα πρέπει να την ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω για το μέλλον για να δημιουργήσουμε μια γνήσια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη να επιδείξουν ρεαλισμό τα κράτη-μέλη στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι και να αποφασίσουμε για το δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε στο μέλλον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Μέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή Συνεροφυλακή και Ακτοφυλακή θα έχει προσωπικό χιλίων προσώπων και 335 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο προϋπολογισμό. Εάν, για παράδειγμα, θέλουμε να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα του οργανισμού με 3.000 υπαλλήλους σε μόνιμη βάση, χρειαζόμαστε 20 με 25 δισεκατομμύρια χείριση των συνόρων. Χρειάζεται 130.000 ε, υπαλλήλους και αντίστοιχο, αντίστοιχο ε, του ετήσιου προπολογισμού της Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, η απόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό θα είναι πολύ νεροφυλακής και ακτοφυλακής. Ενισχύσαμε επίσης και την εντολή της για τις επιστροφές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει όλοι μας ότι η επιστροφή όλων εκείνων που δεν έχουν το δικαίωμα να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία, να εξασφαλίσουμε τη μόνιμη υποστήριξη στις αυξανόμενες προσπάθειες υποδοχής εκείνων που πραγματικά χρειάζονται προστασία. Το θέμα δεν είναι μόνο οι επιστροφές όμως. Αντίστοιχα και, και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία για τους καλή τυπίστη ταξιδεύοντες. Ήδη έχουμε επιτελέσει σημαντική πρόοδο. Το νέο σύστημα ε, εισόδων εξόδων έχει συμφωνηθεί για να ενισχύσουμε τα εφιστάμενα συστήματα όπως είναι το SIS, σύστημα προφόρησης έγκαιρ, το ΕΚΡΙΣ ε, για τα ποινικά μητρώα και ακόμα περισσότερα. Και πάλι αυτό που χρειάζεται είναι να επιτύχουμε ταχεία συμφωνία για τα θέματα αυτά που σας ανέφερε μόλις. Σε μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, 92% των μία για τα θέματα αυτά που σας ανέφερε μόλις. Σε μια πρόσφατη Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, 92% των Ευρωπαίων πολιτών συμφωνούν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μοιράζονται τις προφορίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμούν καταστήσουμε τα συστήματά μας διαλειτουργικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, το σοβαρό έγκλημα και να ε, φυλάξουμε τα σύνορά μας, όπως είπα προηγουμένως. Συνοριοφύλακες, αστυνομικοί, ε, αρχές δικαστικές, αρχές μετανάστευσης θα πρέπει να έχουν ε, μία διεπιφάνεια ενιαία, ένα πόρταλ ε, έρευνας για όλα τα κεντρικά συστήματα. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε λοιπόν, έχουμε πολλά εργαλεία και υλικά για να ενισχύσουμε τερό. για το λόγο αυτό και μετά από συζητήσεις που είχαμε και μαζί σας και με τα κράτη-μέλη πρόκειται να καταθέσουμε την πρότασή μας για μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Εφαρμόζουν τους κανόνες έγκαιρα και όχι μόνο, να συνεργάζονται ε, ε, τη βάση του ιδίου πνεύματος της ίδιας αποστολής και να τους εκπαιδεύσουμε για να γίνουν ένα σώμα συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ε, γνήσια ευρωπαϊκό. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω, αν μου επιτρέπετε, ένα πολύ σημαντικό. Πευθύνουμε έκκληση στο Συμβούλιο να αποφασίσει επιτέλους για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να αποφασίσει να ενταχθούν στην οικογένεια του Σέγγεν. Και φυσικά και η Κροατία αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη χώρα σε τεχνικό επίπεδο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική, να συνεχίσουμε τη συνεργασία για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, συνυπευθυνότητας και εμπιστοσύνης. Παράλληλα, από κοινού θα πρέπει να ενισχύσουμε και να διαφυλάξουμε το και οικονομικά και κοινωνικά και γεωγραφικά. Και το Σέγγεν είναι η εγγύηση μιας γεωγραφικά ενωμένης Ευρώπης που εξασφαλίζει την ενότητα των εθρών μας και των κρατών και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μόφωνα στην Επιτροπή μας με αυτά που είπατε για την ενότητα που χρειάζεται για την ε, ολοκλήρωση του Σέγγεν. Ας περάσουμε τώρα όμως στις... Εκπροσωπείται τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Μόνο για πολιτικό πλήγμα, μίλησε και για οικονομικό πλήγμα και μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό το οικονομικό πλήγμα. Σύνορα. Αυτά που έλεγε η Τάνια. Φανταστείτε ένα Ρουμάνο, ας πούμε, που είναι Ευρωπαίος πολίτης. Με την ίδια έννοια που είναι ο Γερμανός Ευρωπαίος πολίτης πρέπει ας πούμε να περάσει από τέσσερις νοριακούς ελέγχους για να φτάσει στη Γερμανία μέσω της Αυστρίας. Αυτό σημαίνει από τη Βουλγαρία ε, στην Αυστρία. Ε, με ξαναέλεγξαν, γιατί δεν, η, η Βουλγαρία δεν είναι στον χώρο Σέγγεν. Μετά πήγα στη Βουδαπέστη. Εκεί δεν με έλεγξαν γιατί